Good morning, everybody. Dear colleagues, please take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Busy schedule, as usual. Γιατί προχωράει η ώρα και καλό είναι να αρχίσουμε. Έχουμε και ψηφοφορίες, αλλά πρώτα ανακοινώσεις. Αν μου επιτρέπετε. Οι ανακοινώσεις αφορούν ε, της κατεξοδότηση πράξης και τις εκτελεστικές. Η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Βίζα και τα σύνορα, το Ταμείο Συντερικής Ασφάλειας και το ΑΣΥΦ, ε, μάλλον το ΑΜΥΦ, το, Ταμείο για τη Μετανάστευση κτλ. Η ε, Ολομέλεια ε, ψήφισε αντίρρηση σε δύο κατουσιοδότηση πράξεις για αυτά τα δύο θέματα. Τον Οκτώβριο του 2019, στις 15 Οκτωβρίου, ε, λάβαμε δύο νέες κατεξουδότησης πράξεις για το ΑΜΥΒ. Δύο μήνες προθεσμία για να προβάλλουν αντίρρηση το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Several political groups. Διάφορες πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές και δημοκράτες, γκουε, πράσινοι και ρινιού, ε, ζήτησαν το σημείο αυτό να προσθεθεί στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για να ενημερωθούμε ε, επί της ουσίας αυτών των ε, δύο κατεξουδότηση πράξεων και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε δεόντως για την κατάρτιση αυτών των δύο νέων ε, πράξεων. Γι' αυτό προσεκλήθη ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Home για να καταθέσει δύο νέες τις δύο νέες αυτές προτάσεις στι 21 Νοεμβρίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Προηγουμένως θα γίνει τεχνική συνεδρίαση στις 11 Νοεμβρίου με του πολιτικούς συμβούλου. Στη συνέχεια, στις 30 Οκτωβρίου το Κοινοβούλιο έλαβε την εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1585 του 2015 που αφορά τον κατάλογο των υποστηρικτικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλουν ε, πολίτες του ε, Αζερμπαϊτζάν για ε, θεωρήσεις ε, βραχίας διάρκειας. Όλα τα μέλη ΛΥΜΠΕ έλαβαν τα σχετικά γραφά μέσω του newsletter στις 31 Οκτωβρίου. Έχει οριστεί και εσωτερική προθεσμία για αντίρρηση που είναι η 13η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις. Και φυσικά θα πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των προηγουμένων συνεδριάσεων. Ωραία. Εγκρίνονται. Αν δεν διαφωνείτε, θαυμάσαι. Πάμε στην ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική είναι και έχει να κάνει με το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνειροφυλακή και Ακτοφυλακή και την κοινή δράση ε, του Συμβουλίου 98 κάθετος 700 είναι ο αντίστοιχο κανονισμό. για το αντίστοιχο σύστημα. Είναι εδώ η συγκεκριμένη κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα και έχουμε ψηφοφορίες και συμβιβαστικές και χωριστές και μπλοκ. Πρώτον, έχετε όλοι τις κάρτες σας έτοιμες. Είστε έτοιμοι να ψηφίσετε. Η συγγήτρια έχει να πει τίποτα. Όχι. Πάμε αμέσω στη ψηφοφορία. Ωραία. Ψηφίζουμε. On block. Κάποιες συμβαστικές πρώτα που θα πρέπει να ψηφιστούν μαζί. Και αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Αρχίζει, είπα. Ας block. Πέρας. 54, 5 αποχές και μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε τις παραγράφους. Συμβιβαστική στο άρθρο 80. Ε, αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε. Τώρα, η συμβαστική τροπολογία για το άρθρο 80α νέο που καλύπτει τροπολογία 26. Open. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβαστική στο άρθρο 8β νέο που καλύπτει τις τροπολογίες 27 και 58. Αρχίζει ψηφοφορία. Now close. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, στο άρθρο 80 συνέο η συμβαστική που καλύπτει τις τροπολογίες 28, 57, 53 και 61. Αρχίζει ψηφοφορία. Now closed. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Ε, τώρα θα ψηφίσουμε τη συμβιβαστική στο άρθρο 80D. Νέο. Καλύπτει την τροπολογία 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Now closed. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Προχωρούμε στο άρθρο 80 ή νέο ναι, καλύπτει τις τροπολογίες 30, 62 και 68. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πάμε στο συμβιβασμό για το άρθρο 80F νέο. Καλύπτει η τροπολογία 31, 66, 59. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 80D. G, ε, συγγνώμη. Νέο. Καλύπτει την τροπολογία 32 και 72. Αρχίζει ψηφοφορία. G. 80G. Όπως Γρανάδα. 32 και 72. Πέρασε. εγκρίνεται. Συμβιβασμό για το άρθρο 80H. κάλυπτει τις τροπολογίες 33, 34 και 73. Ψηφίζουμε. Αρχίζει ψηφοφορία. Now it's closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα, ο συμβιβασμός στο άρθρο 80J. Νέο που καλύπτει ε, τις 35 και 69. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβιβασμό στο άρθρο 80 και νέο. Καλύπτει την τροπολογία 36. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα προχωρούμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Σε αιτιολογικές σκέψη recital 80. Καλύπτει τη τροπολογία 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Με με μεγάλη διαφορά. Τώρα έχουμε το συμβασμό για την αιτιολογική σκέψη 81β ναι Καλύπτεται η τροπολογία 5 και η 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η ε, αιτιολογική σκέψη 81 C νέα όχι, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Ε, τροπολογία 39. Χωριστά ε, ψηφίζουμε για το συμβιβασμό ε, στην 81B. Χωριστά την 39. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και προχωρούμε στην 81 ΣΥΝΕΑ. Καλύπτεται τροπολογία 638, 41 και 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, αιτιολογική σκέψη 81, ε καλύπτονται οι τροπολογίες 8 και 45 αρχή ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ε, προχωρούμε ε, στο 81F. Ναι. Οι τροπολογίες 9 και 46 καλύπτονται από το συμφωσμό αυτό. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 81G. Ναι. Καλύπτει τις τροπολογίες 10 και 47. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Στο 82 τώρα έχουμε τις τροπολογίες 11 και 48 που καλύπτει η συμβαστική τροπολογία. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα έχουμε τη συμβαστική τροπολογία στην επιλογική σκέψη 101α. 101α, νέο. Ναι. Καλύπτονται οι τροπολογίε 15 και 51. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 113α, νέο και 114. Τροπολογίες 29, 23 συγγνώμη, και 49 καλύπτονται. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε αρχίζει τώρα ηλεκτρονικά και ονομαστικά φυσικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε ως ήθιστε την απόφαση για την εντολή για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, καθώς επίσης και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. Εδώ χρειαζόμαστε απόλυτη ε, πλειοψηφία για να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Μάλιστα, την έχουμε την απόλυτη ε, πλειοψηφία και παραπάνω και με μεγάλη διαφορά εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια κυρία Μετσόλα. Και προχωρούμε. Προχωρούμε με την ημερησία διάταξη χωρίς διακοπή. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν, ησύχως παρακαλώ. Αλλά κυρίως αυτοί που αποχωρούν και αυτοί ησύχως. Let me announce what the following point... Να σας ανακοινώσω το επόμενο σημείο στην Ευρωπαϊκή Διάταξη. Πρόκειται για το σημείο 12 γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Υπόπτη Προστασία των Δεδομένων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία των Δεδομένων για τον αντίκτυπο της νομοθεσίας, της Αμερικανικής νομοθεσίας Cloud, επί του πλασίου προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δεδομένα και τι εντολέ για τη διαπραγμάτευση μια συμφωνία υπευρωπαϊκή ε, Ένωση για τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικέ αποδείξει για δικαστική συνεργασία σε ποινικέ υποθέσει ε, και πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση τη Βουδαπέστη. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε την παρουσίαση του Βόησες Βιεβορόφσκι. Τον ε, καλωσορίζουμε, ο οποίος είναι βοηθός επόπτης ε, του Ευρωπαίου Επόπτη για την Προστασία των Δεδομένων ε, και θα ακούσουμε και τον κύριο Κάρστεν Μπέιν, ε, ο οποίος είναι σύμβουλος πολιτικής στην Γερμανία για την προστασία των δεδομένων και θα ακούσουμε και την παρουσίαση Τιέν Μωρή, νομικού από την ΚΝΙΛ που είναι η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών στη Γαλλία. Ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Βιεβορόφσκη και κατόπιν θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις της νομικής υπηρεσίας, της γνωμοδότησης της νομικής υπηρεσίας που είναι σχετική με το έργο που έχουμε να υλοποιήσουμε προκειμένου να αξιολογήσουμε όπως πρέπει την πρόγνωση αυτής της συμφωνίας ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Έχετε το λόγο, κύριε Διαβαρόσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής. Ε, συλλέγουμε ηλεκτρονικές ε, ψηφοφορίες και από τις άλλες ε, δικαιοδοσίες. Αυτό είναι το θέμα που θα παραμείνει στη μερσία διάταξη αυτής της Επιτροπής ε, για όλη τη θητεία. Αυτό συνδέεται με τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες και με το έργο για το πρόσθετο πρωτόκολλο για τη σύμβαση για το, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο αλλά επίση είναι σημαντικό για τι εσωτερικέ μα συζητήσει για την πρόταση για τι ηλεκτρονικέ αποδείξει. Είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά πιο συγκεκριμένα επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα εμπλέκεται σε διάφορε διαδικασίε για να καταστήσει του κανόνε ε, για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδείξεων και γενικά ηλεκτρονικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά διάφορα ε, ηλεκτρονικά ίχνη διασυνοριακά σε διάφορα φόρα και με διάφορα κράτη, όχι μόνο ευρωπαϊκά κράτη και όχι μόνο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Τον Απρίλιο του 19 εκδώσαμε δύο γνωμοδοτήσεις που θα σας αναφέρω. Σύσταση της Επιτροπής για την διαπραγματευτική εντολή σύναψης Διεθνούς Συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για διασυνοριακή πρόσβαση σε αποδείξεις και τη συμμετοχή της διαπραγματεύσης για το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο για τη σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Και φέτος τον Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Προστασίας Δεδομένων μαζί με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη έδωσαν απάντηση σε αυτή την Επιτροπή για τις επιπλοκές ε, του Cloud Act που υιοθέτησαν οι Ηνωμένε Πολιτείες για το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, για την προστασία των δεδομένων. Χθε, εκδώσαμε μια πρόσθετη γνωμοδότηση που σχολιάζουμε τη σημερινή συζήτηση για την πρόταση ηλεκτρονικών αποδείξεων. Σκοπεύω να επικεντρωθώ σε κάποιες γενικές αρχές στα σχόλιά μου και να ενημερώσω τις απαντήσεις του EDPS, του Ευρωπαίου Απόπτη, στις διάφορες πρωτοβουλίες και σε κάποια συγκεκριμένα σημεία από τη χθεσινή γνωμοδότηση για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι συνάδελφοι από το Συμβούλιο Προστασίας των Δεδομένων έδωσαν κοινή απόνταση για ε, την ε, πράξη Cloud Act και τις επιπτώσεις. Ε, έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του επόπτη από την αρχή και κυρίως για τον Τζουβαλί Μουταρέλη, ο οποίος ε, παρουσίασε την προπτική του ως ε, δικαστής, από δικαστική σκοπιά για το θέμα αυτό. Αναγνωρίζουμε πλήρως ότι οι αρχές, ακόμη και αν ε, ερευνούν εγχώριες υποθέσεις, συχνά πρέπει να ζητήσουν πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε άλλη χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αποτελεσματικούς κανόνες για να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και επίσης ε, βιώσιμες διευθυντήσεις με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή των δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου. Ωστόσο, καταρχήν αυτό είναι το κύριο ζήτημα, το θέμα της δικαιοσύνης και όχι της προστασίας των δεδομένων. Ταυτόχρονα, η συλλογή των αποδείξεων σημαίνει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και εντάσσεται λοιπόν στο πεδίο της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Έτσι λοιπόν έχουμε και θέματα προστασία των δεδομένων και δικαστικά θέματα ταυτόχρονα. Αυτό ενδιαφέρει τις αρχές Προστασία των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία των Δεδομένων. Η συνεργασία με το EDPB και το EDPS ε, δοκίμασε την, ε, δυνατό, την ικανότητα να προσεγγίσουμε τα θέματα που είναι τόσο πολύπλοκα από πολλαπλές σκοπιές και χαίρομαι που θα σας ενημερώσω ότι πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα είναι απολύτως ικανοποιητικό. Γι' αυτό μέχρι τώρα αποφασίσαμε να μην παρεύουμε εμεί ω ε, Ευρωπαίο Επόπτη τα δεδομένων. Ε, αποφασίσαμε να μην εκδώσουμε επίσημη γνωμοδότηση και εκδόθηκε η γνωμοδότησή μα χθε κατόπιν αιτήματο. Το κύριο μήνυμα μας για την όλη συζήτηση είναι ότι η προστασία των δεδομένων δεν εμποδίζει μια αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Τα πρότυπα της προστασίας των δεδομένων, το αντίθετο, θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη και την ακαιρεότητα της απονομής της δικαιοσύνης. Η ουσία των ατομικών δικαιωμάτων δεν εξαφανίζεται τη στιγμή που ο ανακριτής αποφασίζει ότι σε μία ε, ιδιωτική οντότητα, έναν πάροχο τηλεπικοινωνιών, παραδείγματο χάρη, θα πρέπει ο πάροχο αυτό να παραδώσει πληροφορίε σχετικέ με την έρευνα. Η πολυπλοκότητα αυτού του φακέλου προκαλείται κυρίω από το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να οικοδομεί τον κοινό δικαστικό χώρο. Ο κοινό δικαστικό χώρο ε, είναι υποδιαμόρφωση. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ αποκλήσει μεταξύ των διάφορων συστημάτων ε, ποινική δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν, παραδείγματο χάρη, ακόμη παράνομη την άμβλωση και αναγνωρίζεται σοβαρό έγκλημα ε, Παραδείγματο χάρη το θέμα τη ε, προδοσίας μπορεί να ε, διαφέρει στο πώς εκτιμάται στο Παρίσι, στο Τάλιν, αλλά ακόμη και μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελόνης. Κάποια συστήματα ποινικού δικαίου κάνουν διάκριση μεταξύ της προδοσία. χάτης προδοσίας και προδοσίας και μπορεί να προβλέπονται και διαφορετικές ελάχιστες ποινές ε, για τέτοια εγκλήματα. Ε, μπορεί να υπάρχουν ε, κάποιες προβλέψεις στον Εθνικό Ποινικό Κώδικα. Όμω η κατάσταση είναι πολύπλοκη. Δεν υπάρχει, παραδείγματο χάρη, ένα και μόνο ορισμό για το ότι πρόκειται για σοβαρό έγκλημα. Και αρχίσουν να... και υπάρχει διαφοροποίηση ακόμη και εδώ στο Κοινοβούλιο την διαπιστώνουμε. Όμως αυτό είναι σημαντικό από τη σκοπιά της προστασίας των δεδομένων. Ταυτόχρονα έχουμε το εναρμονισμένο πλαίσιο που εφαρμόζεται απευθεία και ανήκει στην πρωτογενή νομοθεσία και είναι η Χάρτα των Θεμελιών Δικαιωμάτων. Και έχουμε και τον DGPR, τον Κανονισμό Προστασία των Δεδομένων, και έχουμε και την Οδηγία για την Αστυνομία, όπω αποκαλείται. Είναι η μόνη οδηγία που εφαρμόζεται από το δευτερογενέ επίπεδο σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. και σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ. Υπάρχουν σημαντικές αναντιστοιχίες στο επίπεδο εναρμόνιση μεταξύ τη απονομή δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τη επιβολή των κανόνων για την προστασία των δεδομένων. Συνεπώ, κάθε φορά που προτείνεται ένα ευρωπαϊκό μέτρο στον τομέα της δικαιοσύνης και της ασφάλειας που θα περιόριζε τα θεμελιώδη δικαιώματα ή που θα παρέμβαινε στα θεμελιώδη δικαιώματα, έχουμε τις ίδιε νομικέ δυσκολίες. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τώρα τις δυσκολίες αυτές πριν να προτείνω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο περιορισμός υπερστολή των δικαιωμάτων μπορεί να είναι νόμιμη μόνο αν γίνει αναλογικά στη δημοκρατικά κράτη και σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μας βοηθά να το αξιολογήσουμε. Εδώ αναφέρομαι και σε άλλες γνωμοδοτήσεις όπως η γνωμοδότηση για το PNR, τους καταλόγους ε, επιβατών. Η πρόταση ηλεκτρονικών αποδείξεων ε, που έχουμε επιτάπητος θα δημιουργήσει την απέτηση η ιδιωτική οντότητα να παραδώσει ευαίσθητα δεδομένα στην δικαστική αρχή σε άλλη δικαιοδοσία. Όσο λαμβάνει η χώρα σε ένα σύστημα που δεν έχει οικοδομηθεί από την αρχή, το αντίκτυπο αυτού του, ε, του μέσου θα ήταν ε, ενδυνάμει σημαντικό σε ό,τι αφορά την ε, περιστολή των δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας. Όλα όμως εξαρτώνται από την ανάλογη υπόθεση και μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανά υπόθεση. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τον ψύχη ψηλά σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες για να ε, δούμε ένα παράδειγμα. Παραδείγματο χάρη, πάρτε ένα κρατό μέλο που γνωρίζετε το λιγότερο και προσπαθήστε να φανταστείτε ποιο ε, είναι ο κατάλογο των αρχών τη χώρα αυτή που έχουν τις προϋποθέσεις ε, για να ζητήσουν τα δικά σας δεδομένα από έναν πάροχο. Παροχή υπηρεσιών ε, και προσπαθήστε να δείτε ποια είναι τα σοβαρά εγκλήματα στο κράτος προς το οποίο η αίτηση και να ε, θέλετε έναν ενδιάμεσο πάροχο παροχής υπηρεσιών ή πιστεύετε ένας πάροχος παροχής υπηρεσιών θα ξέρει όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θέλετε ο πάροχος παροχής υπηρεσιών να απαντήσει μόνος του ή θα προτιμούσατε ο δικαστής στη χώρα σας να βοηθήσει αυτόν τον πάροχο. Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τα δεδομένα συναλλαγών, φανταστείτε ότι οι πληροφορίες με το ποιον θα τις επαφή και πού βρισκόσασταν είναι μέρος αυτών των δεδομένων. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να είναι ο ιδιωτικός πάροχος, πραγματος χάρη, ε, ο πάροχο ίντερνετ για να κρίνει ποια είναι η αναλογικότητα και η νομιμότητα του αιτήματο για την παροχή προσωπικών δεδομένων ε, στη δικαστική αρχή μια αλλοδαπής δικαιοδοσία. Ε, δεν έχει σημασία τώρα εδώ αν έχουμε κατά νου κράτο Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτη χώρα. Εμείς στην γνωμοδότησή μας συμβουλεύουμε ε, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την επιβολή των κανόνων και θα πρέπει να είναι συνεκτική με τους υφιστάμενους ε, όρους της κατηγορίας της Ευρωπαϊκής. Συγγνώμη με τις ε, κατηγορίες των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξει και βελτίωση σε ό,τι αφορά ε, τους όρους του content data και του transactional data και δίνουμε συμβουλή να, τροποποιηθούν προ... να τροποποιηθεί η πρόταση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι δυνατόν η επάρξη εμπλοκή του δικαστή και στις δύο δικαιοδοσίες και του κράτους έκδοσης και ε, του κράτους επιβολής του νόμου. Φυσικά η εταιρεία στο κράτος της επιβολής ε, θα πρέπει ε, να δικαιούται να ζητήσει δικαστικό έλεγχο και δικαστική βοήθεια. Να γνωρίζουμε ότι ε, υπάρχουν ε, κάποιες καθυστερήσεις όπως έχουμε στην αμοιβαία συνδρομή και προσπαθούμε να βρούμε λύση. Όμως, είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα που να είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και ταχύ. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του είδους ε, του αδικήματος ε, για το οποία μπορεί να εκδοθούν ευρωπαϊκά εντάλματα ε, για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ε, και ε, της, του αιτήματο συνένεσης του υποκειμένου. Επίσης θα πρέπει όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων να είναι ασφαλείς. Ο Ευρωπαίος Επόπτης θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, θα προσπαθήσει να αξιολογήσει τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Για να ολοκληρώσω, πρόκειται λοιπόν ένα σημαντικό σταυροδρόμι υπερταξύ των αναγκών της δικαιοσύνης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων. Ελπίζουμε ότι η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Έργων Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Πόπτη θα βοηθήσει να κατανοήσουμε όλες τις πτυχές αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ευχαριστώ και εγώ. Γνωρίζετε πόσο μας ενδιαφέρουν οι εκθέσεις του επόπτη προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων όταν πρόκειται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και της ιδιωτικότητάς τους. Είναι ανησυχητικές οι ε, νομικές εξελίξεις Γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε και τον κύριο Κάνστεντένα ε, για να συμπληρώσουμε τις γνώσεις μας για ε, τα θέματα αυτά. Είναι από το Γερμανό επόπτη προστασίας δεδομένων. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, ο κύριος Ντένεν. Καλημέρα σας, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και από πλευρά του Γερμανού Επόπτη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων θα θέλαμε να σα ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση που μα απευθύνεται και την ευκαιρία που έχουμε σήμερα ε, να συζητήσουμε και να απαντήσουμε. Ε, αυτή είναι η βάση της ε, παρουσίασής μας. Είχαμε ξανάρθει στην Επιτροπή, μάλλον η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ η προηγούμενη μας είχε ζητήσει να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις της Αμερικανικής νομοθεσίας Cloud Act στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Πριν προσπαθήσω να συνοψίσω ε, τα συμπεράσματά θέλω να προεξοφλήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή η εκτίμηση είναι μια αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε σε αυτό το θέμα που είναι τόσο περίπλοκο και θα ετοιμάσουμε πλήρη γνωμοδότηση για το επόμενο έτος για θέματα αυτά και άλλα σχετικά. Ε, και κατά δεύτερο λόγο, ε, η απάντηση που σας δώσαμε αφορά ένα ειδικό σενάριο σε περίπτωση που υπάρχει ένταλμα από μια διοκτική αρχή σε μια ποινική έρευνα, αμερικανική αρχή. Τα συμπεράσματά μας λοιπόν ε, είναι διαφορετικά και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, είναι διαφορετικό το αίτημα και αν άλλη αρχή που εμπίπτει σε άλλο κλάδο του δικαίου το ζητήσει. Ε, αφού λοιπόν τα προεξόφλησα αυτά τα δύο, θέλω να σας παρουσιάσω το βασικό μας συμπέρασμα. Ε, τι λέμε. Εάν δεν αναγνωρίζεται ε, βάση ε, διεθνού συμφωνία το αίτημα και με την επιφύλαξη κάποιων ειδικών ε, περιπτώσεων για τα ζωτικά συμφέροντα του ενδιαφερομένου, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να προβούμε ε, με βεβαιότητα ε, σε αποκάλυψη των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση ε, θα δημιουργηθεί σύγκρουση. Και προσπαθούμε στην υπόλοιπη επιστολή να προτείνουμε κάποια μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορες διεθνείς συμφωνίες. Η πρώτη είναι μια νέα γενιά συμφωνιών αμοιβαία δικαστικής συνδρομής. Ε, αυτό είναι ένας τρόπος και πιο γρήγορος ε, και πιο ειδικό για να έχει ασφαλιστικέ δικλείδε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά δεύτερο λόγο, αναφερόμαστε σε συμφωνίε όπω είναι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ που ήδη είναι υποδιαπραγμάτευση. Θα μπορούσε να λύσει αυτό το θέμα. Αυτό θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αν είναι αρκετές οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων. Γιατί νομίζουμε ότι θα μπορούσε αυτό να λύσει τις συγκρούσεις και να επιφέρει μια νομική ασφάλεια που θέλουμε όλοι. Ε, επίσης θέλω να τονίσω άλλα δύο σημεία. Εκφράζουμε μεγάλη προτίμηση στο να είναι η συμφωνία όχι διμερής αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών και όχι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και μονομένων κρατών μελών τη Ένωση. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι ανάγκη να υπάρχει συνέπεια και συνοχή ε, στη στάση μα. Τι εννοώ. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα υπάρχει εδώ πιο μεγάλη ευελιξία, ελαστικότητα ε, σε σχέση με τα αιτήματα ε, που γίνονται ε, από διοκτικές αρχές των ΗΠΑ σε άλλες διοκτικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταματώ εδώ και θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ετιέν Μωρή. Thank Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τον Ετιέν Μωρή που είναι νομικός σύμβουλος ε, του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων στην ε, ΚΝΙΛ, ε, στη Γαλλία. Έχουμε και άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό και θα ακούσουμε την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίπτωση της εφαρμογής της Αμερικανικής Νομοθεσίας Cloud Act στην εντολή μας για τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες για τη σχετική συμφωνία για τη ευκόλυνση πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για όλους μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μωρή. Merci, Monsieur σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Μετά από τις, τα γενικά συμπεράσματα, καθώς επίσης και τις συστάσεις που ο προελίσσης συνάδελφος ε, σας ε, ανέφερε, θα ήθελα να αναφερθώ στο παράρτημα της, επιτροπής, ε, της επιστολής συγγνώμη, που εστάλει στην Επιτροπή σας. Θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση βασιζόμενο σε δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα τις επιπτώσεις του Cloud Act ή σε ε, τη διασυνορική πρόσβαση στα δεδομένα και δεύτερον στην ε, διάδραση ανάμεσα στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως το RGPD ε, και το Cloud Act. Ε, όσον αφορά τις διατάξεις ε, του Cloud Act της 23ης Μαρτίου 2017, όπως γνωρίζετε αυτό, αυτή η νομοθεσία αποτέλεσε συνέχεια πολλών στοιχείων τα οποία συζητήθηκαν στην διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως δε μετά από την υιοθέτησή της ακυρώνεται η υπόθεση Microsoft για την οποία αναμένεται το απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Ε, το Cloud Act ε, αναφέρει ότι οι Αμερικανικές αρχές μπορούν να υποχρεώσουν ε, τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών κτλ. να δώσουν πρόσβαση στις ΗΠΑ σε στοιχεία αποθηκευμένα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, η νομοθεσία αυτή αναφέρεται, αναφέρει ότι μπορούν αντίστοιχα και οι χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών να ζητήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση σε στοιχεία που είναι εκεί αποθηκευμένα ε, με την προϋπόθεση να είναι ε, οι λεγόμενες επιλέξιμες. Ε, για την δική μας επιτροπή η Cloud Act ε, καθιερώνει ένα σύστημα το οποίο ξεπερνά τη συμβάση δικαστικής ε, συνδρομής. Ε, τροποποιεί λοιπόν την Stored Communication Act και υποχρεώνει εφ' εξής τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής Κοιτάξτε, ε, μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, λέει ο Πρόεδρο, ε, και επομένως οι διερμηνείς έχουν πρόβλημα. Ε, υποχρεώνει λοιπόν τους ε, παρόχους που ανέφερα προηγουμένως να διατηρούν και να προωθούν το περιεχόμενο είτε μια επικοινωνία, είτε μια ηλεκτρονική επικοινωνία, είτε οποιαδήποτε καταγραφή ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά ένα πελάτη ή ένα μέλο το οποίο κατέχει, διακατέχει ή ελέγχει αυτός ο πάροχος, ε, είτε πρόκειται για το εσωτερικό είτε πρόκειται για το ε, ε, εξωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό ε, να ε, πούμε ότι η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή μας στα πλαίσια αυτά έχει καταγράψει ότι το Cloud Act δεν επιτρέπει την, την μαζική συλλογή και την συστηματική προώθηση των προσωπικών στοιχείων, αλλά θέλει να κάνει μια διευκρίνηση όσον αφορά την εδαφική ισχύ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι έχουμε αφενός την πρόσβαση ε, των δεδομένων περιεχομένου, ε, πρόσβαση στα μεταδεδομένα επί τη βάση μιας ε, επιβολής ή ακόμα και σε περίπτωση κατάσχεσης και τέλος τηλεφωνικών παρακολουθήσεων σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος έχει ε, ε, βρίσκεται σε μια χώρα η οποία διαθέτει ήδη συμφωνία ε, εκτελεστική με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια τελευταία διάταξη που είναι σημαντική αναφέρει ότι δεν θα μπορούσαν οι πάροχοι να μεταφέρουν τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται προστατευμένα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ε, εάν, υπάρχει μια χώρα η οποία δεν ε, ε, συμφωνεί με την πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει εκτελεστική συμφωνία και δεν βρίσκεται επομένω μεταξύ των επιλεξίμων χωρών, μπορεί να μην προσφύγει σε τον μηχανισμό επίλυσης που προβλέπεται από την Cloud Act. Αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μονάχα σε περίπτωση χωρών που διαθέτουν ήδη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, μέχρι τώρα δεν έχει υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα το οποίο ετέθη, ε, ε, το, η Ευρωπαϊκή μας ε, Επιτροπή Προστασίας έχει καταγράψει το εξής. Μια ευρωπαϊκή ε, εταιρεία ή ένας ευρωπαϊκός πάροχος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να ε, ε, συμμορφωθεί με την Cloud Act. Αναφέρεται αυτή σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο ενός παρόχου. Υπάρχει όμως η περίπτωση και εδώ παραθέτω το RGPD, ένας υπεύθυνος διαχείρισης ή ένας υπεργολάβος να χρειαστεί συγκεκριμένη εντολή έτσι ώστε να δώσει τα στοιχεία αυτά. Στο άρθρο 48 του RGPD αναφέρεται ότι οποιαδήποτε απόφαση ε, ε, ε, κάποιας νομικής υπηρεσίας ή κάποιας διοικητικής αρχής μιας τρίτης χώρας που ε, ζητά από τον υπεύθυνο διαχείρισης ή τον υπεργολάβο να μεταφέρει ή να διαδώσει στοιχεία προσωπικού ε, περιεχομένου δεν μπορεί να αναγνωριστεί ή δεν μπορεί να γίνει εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο παρά μόνο εάν βασίζεται σε διεθνή συμφωνία όπως αυτή της δικαστικής συνδρομής. Με άλλα λόγια, το άρθρο 48 καθορίζει σαφώς ότι για να δώσει ε, πρόσβαση ή για να να παράσχει αυτά τα στοιχεία ε, μια αρχή θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπογράψει μια συμφωνία αντίστοιχη της Σύμβασης Δικαστικής Συνδρομής. Στην προκείμενη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή του Cloud Act, ε, ε, μια ένα αμερικανικό αίτημα το οποίο θα αποσταλεί εκτός των παραδοσιακών διάβλων της δικαστικής συνδρομής δεν μπορεί να γίνει εκτελεστή. Το Κομιτέ Ευρωπαίο θεωρεί ότι μια και δεν υπάρχει εφαρμοστική διεθνή συμφωνία ε, ε, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη νομική βάση ε, σύμφωνα με το RGPD, μια τέτοια, ένα τέτοιο αμερικανικό αίτημα δεν μπορεί να βασιστεί εις την νομιμότητά του. Και επομένως, όταν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, ε, όταν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες μπορούν να απορρίψουν το αίτημα ε, οι εταιρείε και να Ε, να αρνηθούν γιατί ε, εάν δώσουν τα στοιχεία αυτά από τη μία πλευρά ε, θα έχουν αντίθεση σε σχέση με την, το αίτημα των Αμερικανικών αρχών και από την άλλη πλευρά θα έχουν παραβιάσει την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την μετάδοση στοιχείων προσωπικών, προσωπικού χαρακτήρα. Ε, και οπωσδήποτε ε, ε, λαμβάνονται υπόψη και όλα τα στοιχεία αυτά που αναφέρονται είναι υπό την αίρεση άλλων στοιχείων και διατάξεων που προβλέπονται από το RGPD. Αναφέρομαι κυρίως ε, εις ε, ε, στο, στην πλησίωση της μη μετάδοσης εκτός του εδάφους Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχείων προσωπικών δεδομένων. Η πλαισίωση της δυνατότητας μεταφοράς των στοιχείων αναλύεται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται δηλαδή ακόμα υπό ανάλυση. θα ήθελα όμως τελειώνοντας, παρότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται... Ε, στο αίτημα των Αμερικανικών αρχών. Ε, σε αυτή την περίπτωση και αν υπάρχει αίτημα από πλευράς Αμερικανικών αρχών βρισκόμαστε στην περίπτωση άμεσης σχέσης ανάμεσα σε ε, αρχές άλλου κράτους και τις, τους διαχειριστές και παρόχους υπηρεσιών. Αλλά δεν υπάρχει στην προκείμενη περίπτωση καμία προστασία όσον αφορά το, νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει αυτήν την ε, σχέση. Επίσης, μια ε, επιχείρηση η οποία βρίσκεται στις, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομική βάση έτσι ώστε να προωθήσει, να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία ε, καθότι υπερέχει ε, η αρχή της προστασίας του δικαιώματος δηλαδή του ατόμου να προστατέψει τα προσωπικά του στοιχεία. Ε, μετά από πρόταση του κανονισμού για την πρόσβαση ε, σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, ε, η προστασία των στοιχείων πρέπει να είναι ε, όσο πιο αποτελεσματική γίνεται και όσο πιο αποτελεσματικά προβλέπεται από τις εθνικές αρχές. Ε, και ε, οπωσδήποτε υπάρχουν και όλα τα εχέγγυα, εφαρμόζονται μάλλον όλα τα εχέγγυα τα οποία προβλέπονται στις συμβάσει δικαστικής ε, συνδρομής. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη διεθνής συμφωνία και υπό την αίρεση ύπαρξης εξαιρετικών προϋποθέσεων δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης της νομιμότητας του αιτήματο από πλευράς των Αμερικανικών αρχών. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η δική μας Επιτροπή ε, αναφέρει ότι ε, οπωσδήποτε υπάρχει το νομιμοποιημένο αίτημα για βελτίωση της συνεργασίας και καθίσταται αναγκαία η καλύτερη διεθνή συνεργασία και οπωσδήποτε περαιτέρω συζήτηση ε, για το θέμα της ανταλλαγής ή παροχής στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα προς τις Αμερικανικές αρχές. Θα πρέπει να βρεθεί μια συμφωνία η οποία και θα καλύπτει τις ε, προσωπικές ελευθερίες των ατόμων και θα καλύπτει τις διεθνείς ε, απαιτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μωρή. Να περάσουμε τώρα στην νομική υπηρεσία. Ας έχουμε ε, κατά νου της 21 Φεβρουαρίου ζήτησε η Επιτροπή μας ε, μία νομική γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καταρχήν, ε, για τον αντίκτυπο της εφαρμογής ε, της Συμφωνίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείες για την εξοεδαφική ισχύ του εντάλματος και σε σχέση με το Cloud Act και δεύτερον το είναι εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε για αυτή τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να είναι συμβατά με τις ε, ουσιαστικέ νομικές εγγυησει που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς συμφωνίες έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή η πρωτογενής και δευτερογενής νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα που διακυβεύεται εδώ. Για να ακούσουμε την έκθεση της νομικής υπηρεσίας. Ο κύριος Ντάνιελ Βάριν έχει το λόγο για τα επόμενα δέκα λεπτά και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στους βουλευτές για να συζητήσουμε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Επιτροπή σας ε, πράγματι ζήτησε μια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία στο θέμα της νομοθεσίας που θετήθηκε το Μάρτιο του 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απεσαφήνιση της νόμιμης χρήσης των δεδομένων που έχουμε στον νόμο Cloud, Cloud Act όπως ε, τον αποκαλούμε και αφετέρου για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να επιτραπεί μέσω του Συμβουλίου η έναρξη διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένε Πολιτείε προκειμένου να υπάρχει μια συμφωνία για ε, την διασυνορική ανταλλαγή στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας ε, ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται από τους ε, ηλεκτρονικούς παρόχους, τους παρόχους παροχής υπηρεσιών. Έρχομαι σε ένα κύριο σημείο της γνωμοδότησης. Καταρχήν για το Cloud Act. Η Επιτροπή σας ε, αναρωτιόταν για τα αποτελέσματα του Cloud Act ε, δεδομένης ε, της εξοεδαφικής συνιστώσας ε, στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Καταρχήν, η νομική υπηρεσία διευκρίνησε το πόσο εκτείνεται η εξοδαφικότητα του Cloud Act. Ε, ε, πράγματι, έχουμε ένα πεδίο εφαρμογή ε, που υπερβαίνει την επικράτεια των ΗΠΑ, καθώ θέτει ότι οι πάροχοι ηλεκτρονικών περιουσιών δεσμεύονται υποχρεώσει που προβλέπονται από την νομοθεσία σε ό,τι αφορά την αποκάλυψη των πληροφοριών που κατέχουν, είτε είναι αποθηκευμένε είτε όχι αυτέ οι πληροφορίε, στην επικράτεια των ΗΠΑ. Έτσι, λοιπόν, σε, με στοχεύουν σε στοιχεία που μπορεί να έχουν αποδικευτεί είτε εντός είτε εκτός της επικράτειας των ΗΠΑ. Αυτή η εξοεδαφικότητα της Αμερικανικής νομοθεσίας ε, δεν ε, μειώνεται παρά από την απέτηση οι κατασταλτικές αρχές να μπορούν να στείλουν αιτήματα ε, στους παρόχους που υπόκειται στην Αμερικανική δικαιοδοσία. Όμως η έννοια αυτή μένει αρκετά αόριστη ε, δηλαδή το να υπόκειται στην ε, αμερικανική δικαιοδοσία και μπορεί να έχουμε μια εκτεταμένη ερμηνεία από την πλευρά της αμερικανικής δικαιοδοσίας και εν δυνάμει ε, σκοπε, στοχεύει σε πάρα πολλούς παρόχους παροχής υπηρεσιών που θα είχαν έναν χαλαρό σύνδεσμο πάνω κάτω με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Για να αξιολογήσουμε τις συνέπειες αυτής της εξοδαφικότητας θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων του 2016, GDPR, Επίσης ε, έχει και αυτός εξοδαφική, εξοδαφικό πεδίο εφαρμογή στο GDPR βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ε, εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ε, που γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ενός υπεύθυνου επεξεργασίας στο έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επεξεργασία αυτή γίνεται είτε εντός είτε εκτός της Ένωσης και βάσει του άρθρου παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού αυτό εφαρμόζεται επίση ισχύ και σε ορισμένε περιπτώσει για την επεξεργασία των δεδομένων ατόμων που βρίσκονται εντό τη επικράτεια τη Ένωση από έναν υπεύθυνο επεξεργασία που αυτό δεν είναι εγκατεστημένο στην Ένωση. εδώ έχουμε λοιπόν και την πτυχή τη εξοεδαφικότητα του GDPR και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή η διάταξη στοχεύει όχι μόνο σε Ευρωπαίους πολίτες αλλά σε όλα τα άτομα που βρίσκονται στην επικράτεια της Ένωσης με οποιαδήποτε ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα στα δεδομένα του Cloud Act και του GDPR, ένας πάροχος μπορεί να βρεθεί σε μία κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει αντιφατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Αμερικανική νομοθεσία ΦΕΝΟΣ και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία φετέρου, τις οποίες υπόκειται. Γνωρίζοντας ε, αυτή την επιθανή σύγκρουση της νομοθεσίας, ε, οι Αμερικανοί έχουν προβλέψει μια δικλίδα. Έτσι, ο πάροχος υπηρεσιών ε, θα μπορεί να απαλλαχθεί από το να απαντήσει σε ένα αίτημα αποκάλυψης από τους καταστατικούς μηχανισμούς, αν αυτό το αίτημα, αν αυτή η αποκάλυψη, θα οδηγούσε στο να παραβιάσει τον νόμο κάποιας αλλοδαπής κυβέρνησης η κυβέρνηση με την οποία οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έχουν συνάψει διμερή συμφωνία, δηλαδή εκτελεστική συμφωνία που διέπει τη διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά υποδεκτικά στοιχεία. Ε, το συμπέρασμα της η σύναψη τέτοιων συμφωνιών προβλέπεται από το ίδιο το Cloud Act και ε, ο σκοπός είναι να αντικαταστήσουν τη σχέση τη, μάλλον ε, τη διαδικασία της αμοιβές νομικής συνδρομής ε, που μέχρι τώρα έδιεπε τις σχέσεις μεταξύ κρατών σε ό,τι αφορά την απόκτηση αποδείξεων από το εξωτερικό γνωρίζοντα ότι οι διαδικασίες, αυτές οι διαδικασίες αμοιβαίας νομικής συνδρομής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες ε, και καθυστερούν και μάλιστα η πρώτη από αυτές τις συμφωνίες υλοποιήθηκε μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών και μια τέτοια συμφωνία μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτη πρότεινε να θέσουμε από διαπραγματεύσει, όπω θα δείτε στο δεύτερο μέρο των παρατηρήσεων. Αυτέ οι συμφωνίε θα επιτρέψουν την διασυνοριακή ε, δημοσιοποίηση δεδομένων που έχουν Αμερικανοί πάροχοι που ε, τώρα δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Είναι αδύνατο. Η νομική υπηρεσία επίση υπογράμμισε τα όρια τη ασφαλιστική δικλίδα που προβλέπεται από τον Cloud Act. Καταρχήν, έχουμε την αναγκαιότητα να υπάρχει εκτελεστική συμφωνία για να μπορεί να ελοπιθεί, όπως είδαμε. Εξάλλου, η υποχρέωση του να υπάρχει πρώτερη δικαστικό έντελμα για την ε, αποκαλύψη δεν αφορά παρά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ε, επικοινωνίας ε, που έχει στη διάθεσή του πάροχος και όχι άλλες ενδεχόμενες πληροφορίες που μπορεί να διαθέτει ο πάροχος, τα μεταδεδομένα ενώ αυτά τα μεταδεδομένα θεωρούνται επίσης ευαίσθητα δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, σε σχέση με την νομοθεσία της προστασία των δεδομένων. Και η νομική υπηρεσία έχει υποστηρίξει ότι η Αμερικανική δικαιοδοσία είναι αρμόδια να καθορίσει αν η αποκάλυψη που ζητείται από τις Αμερικανικές αρχές θα οδηγούσε ή όχι στον πάροχο των υπηρεσιών στο να παραβιάσει την νομοθεσία ενός τρίτου κράτους. Δηλαδή, η αμερικανική δικαιοδοσία ουσιαστικά θα ερμηνεύσει το λοδοποδίκαιο. Σε σχέση τώρα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συγκεκριμένα το GDPR, η νομική υπηρεσία υπενθύμησε ότι πάροχοι υπηρεσιών που θα μπορούσαν μέσω της εφαρμογή του Cloud Act θα έπρεπε να αποκαλύψουν δεδομένα που κατέχουν στην Ευρώπη. Αν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του GDPR, ε, πρέπει να σεβαστούν τις διατάξεις του σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων προ τρίτες χώρε ενώ αν ε, υπάρχει απουσία ε, των ε, κατάλληλων εγκυρήσεων και υπό την επιφύλαξη των παρεκκλήσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπεται στο άρθρο 49 του κανονισμού, που θα πρέπει να ερμηνευτεί αυστηρά, τα αιτήματα διαβίβασης ε, από την αρχή τρίτης χώρας ε, δεν μπορούν ε, να γίνουν εκτελεστά παρά αν υπάρχει διεθνής συμφωνία όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του GDPR. Ας περάσουμε τώρα στη σύσταση της Επιτροπής για να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη σύνοψη συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ. Υπό την έννοια αυτή, κυρίω έχουμε τις ουσιαστικέ δικαστικές ε, εγγυήσει ε, που θα πρέπει να γίνουν σεβαστές από την ε, μελλοντική συμφωνία σε σχέση με το πρωτογενές και το δευτερογενές δίκαιο. Αυτή είναι η ερώτηση τη Επιτροπής σα. Εδώ θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι κάθε διεθνής, ε, όπως κάθε διεθνή συμφωνία και συμφωνία με τη ΣΥΠΑ δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αντίκειται στις δικές μας συνθήκες και στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Κομισιόν υπενθύμησε στη σασί της αυτή η συμφωνία θα πρέπει να επιτρέψει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γενικών αρχών της Ένωσης που καθιερώνονται στα κείμενα. Αν ε, ε, έχουμε πολλά θεμελιώδη δικαιώματα που μπορεί να, πλη, να θυγούν από την συμφωνία αυτή. Υπογραμμίστηκε επίση ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφο 1 τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κάθε περιστολή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζεται από εκεί πρέπει να προβλέπεται αφενό από τον νόμο και να σέβεται το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτού του δικαίου. Ε, με βάση τη αρχή τη αναλογικότητα, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να είναι απαραίτητοι και να απαντούν σε στόχου γενικού συμφέροντο που αναγνωρίζονται από την Ένωση. Υπό την έννοια αυτή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ήδη ότι ε, η δυνατότητα να διασφαλίσουμε το γενικό συμφέρον αποκρίνεται σε ένα τέτοιο στόχο ε, που μπορεί να αιτιολογηθεί ακόμη και από σοβαρέ ε, παρεμβολέ του δικαιώματο τη ιδιωτική ζωή και τη προστασία προσωπικών δεδομένων, όπω αναγνωρίζεται από τη Χάρτα. Ε, τώρα πρέπει να δούμε αν οι άλλες προϋποθέσεις του άρθρου 52 θα πληρούνται, δηλαδή σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα της ε, περιστολής των δικαιωμάτων από τη μελλοντική συμφωνία. Εδώ η αναλογικότητα αυτή γίνεται πιο εύκολα σεβαστή από μέτρα που έχουν ε, περιορισμένο αντίκτυπο στο δίκαιο αυτό, δηλαδή να είναι κάτι εντελώς απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο στόχο και που συνοδεύονται και από ε, μέσα, μέτρα διασφάλισης. Ε, θα είναι δυνατό βέβαια αυτό να το δούμε μόνο όταν διαθέτουμε το κείμενο της συμφωνίας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά το παράγωγο δίκαιο της Ένωσης, μια διεθνή συμφωνία, υπερισχύει αυτού και μπορεί να υπάρχουν παρεκκλήσεις, όμως θα έπρεπε να τροποποιηθούν νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να μην υπάρχει αντίφαση με το εσωτερικό δίκαιο. Δεδομένων αυτών των παρατηρήσεων και στο στάδιο αυτό η νομική υπηρεσία ε, παρουσιάζει κάποια στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει η μελλοντική συμφωνία για να συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης. Θα βρείτε τα διάφορα στοιχεία στην γνωμοδότηση, θα αναφέρω μόνο ένα εδώ για να απαντήσω στις ανησυχίε ε, που εκφράστηκαν από τον κύριο και μάλλον συμφωνήσω με τις ανησυχίε ότι είναι το πώ ορίζονται ε, τα αδικήματα, παραδείγματο χάρη για τα οποία ζητείται η παροχή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Λοιπόν, για να κλείσουμε, αν η Επιτροπή έχει αναφέρει ήδη αρκετά στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία και αν τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή είμαστε απλά στο στάδιο των προθέσεων και ε, θα πρέπει να δούμε το κείμενο τη διαπραγμάτευση για να δούμε αν αυτό θα προστατεύει πράγματι τα θεμελιώδη δικαιώματα που καθεγρώνονται στη χάρτα και αν θα είναι συμβατό με το παράγωγο δίκαιο τη Ένωση. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Ε, την Αμική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρχίζει η συζήτηση. Σας παρακαλώ, έχετε υπόψη ότι έχουμε άλλα δύο ε, θέματα στην σημερινή ημερήσια διάταξη, πολύ σημαντικά. Ε, έχουμε συζήτηση για το δικαίωμα στη λύθη και μετά έχουμε και κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ στις 11.30 για τελευταίο σημείο του πρωινού. Παρακαλώ να το θυμάστε αυτό, γιατί έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Και καλά κάνουν. Ένα λεπτό όμως ο καθένας για να προλάβουμε. to refrain yourself to... Παρακαλώ προσπαθήστε να περιοριστείτε σε ερωτήσεις. Αν θέλετε και προς την νομική υπηρεσία και προς τους ομιλητές μας. Έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες όμως και παρακαλώ να κάνετε ερωτήσεις. Ε, ωραία. Ο κύριος Ράντεφ πρώτος. Αντιπρόεδρός μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Ακούμε ε, τις παρουσιάσεις ε, των εμπειρογνωμών ε, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για τη δικαστική συνεργασία στο ποινικό ε, δίκαιο. Η συμφωνία αυτή θα βελτιώσει και τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική ασφάλεια. Ε, θα δώσει ένα καλύτερο και ταχύτερο τρόπο εντοπισμού, ανείχνευσης και απάντησης ε, στις τρομοκρατικές απειλές εκατέρωθεν του Ατλαντικού. Ωστόσο, χρειαζόμαστε ασφαλιστικές δικλείδες για τα δικονομικά δικαιώματα ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες που εργάζονται και στις δύο δικαιοδοσίες. Ε, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων προτείνει να ε, προχωρήσουμε ε, σε συμφωνία αμοιβαιότητας και μη διάκρισεων. Ποια είναι όμως τα συγκεκριμένα μέτρα που προτείνετε εσείς ε, για να εγγυηθούμε αυτή την αμοιβαιότητα. Η νομική υπηρεσία στην γνωμοδότησή της εκφράζει ανησυχία ότι η απόφαση για την εντολή αποκάλυψης των Ηνωμένων Πολιτειών που ενδεχομένως να παραβιάζει το δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών μελών αφήνεται στα χέρια των Αμερικανικών δικαστηρίων. Τι λύση μπορούμε να βρούμε γι' αυτό. Κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι του πάνελ. Θα επικεντρωθώ σε μια-δυο επιπλέον ερωτήσεις. Ε, για να είμαστε ε, σύμμορφοι με το ε, GDPR χρειάζεται να έχουμε διεθνείς συμφωνίες. Εκτός αυτού όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε ε, το σύστημα ε, ανταλλαγής δεδομένων που ήδη υπάρχει. Έχουμε και διμερή συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που συνδέεται με τις ε, υποχρεώσεις των εταιρεών για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ε, ασπίδα προστασίας ιδιωτικής ζωής της αντίστοιχη αμερικανικής νομοθεσίας, Privacy Shield. Έχω ειδικές ερωτήσεις και για τους ομιλητές αλλά και για την νομική υπηρεσία. Ε, η νομοθεσία cloud των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δύο τμήματα και έχοντα υπόψη και τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε εξασφαλίσει σε όλε τι περιπτώσει η συμφωνία αυτή ε, να ε, κυριαρχεί επί του πρώτου τμήματος του Cloud Act, ε, όπου προβλέπεται άμεση πρόσβαση στα δεδομένα. Ή μήπω αυτό το πρώτο τμήμα παρακάμψει όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες συμφωνίες και προβλέπεται τίποτα για την μελλοντική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ΗΠΑ και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή τη σύγκρουση. Δεύτερη ερώτηση προς την νομική υπηρεσία. Ισχύει ότι η συμφωνία όταν έρθει Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών θα εμποδίζει τα κράτη-μέλη να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες. Και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών νομίζω είναι πολύ σημαντικό νομικό ζήτημα αυτό. Θα είναι εκτελεστική συμφωνία, δηλαδή δεν θα χρειαστεί ε, κύρωση από το Κογκρέσο ή θα είναι μια κανονική διεθνή συμφωνία όπου χρειάζεται η κύρωση του Κογκρέσου. Επίσης θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για το αίτημα ε, τις απαιτήσει για προδικαστική έγκριση. Δεν το βλέπω να υπάρχει αυτό στην ε, συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Τι γίνεται στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να ε, συμπεριλαμβάνεται εκεί. Και το, ε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσχωρήσει στο GDPR και δεσμεύεται από τον κανονισμό αυτό. Η κυρία Νετβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους τρεις κυρίους του πάνελ για τις πάρα πολύ λεπτομερείς εισαγωγές τους. Θα ήθελα να κάνω κάποια γενικά σχόλια για τη διαδικασία και ο συνάδελφός μου περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχάς, διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη ε, τα όσα λένε οι εμπειρογνώμονες, όπως ε, συνήθως κάνει και, έκανε και στο παρελθόν. Τους αγνοεί. Θέλει, λέει, τα ευρωπαϊκά στοιχεία, τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, ε, για να προχωρήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Μα είμαστε ήδη στο δεύτερο γύρο. Καταπληκτικά πράγματα. Ε, και εσείς τονίσατε πάρα πολύ που υπάρχουν τα νομικά ε, προβλήματα και παραθυράκια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρακαλώ αυτό να γραφτεί στα πρακτικά, εσκεμένα και εγνώση της διαπραγματεύεται με βάση ε, λάθος εντολή. Ξέρουν ότι δεν είναι αεροστεγές αυτό από νομικής πλευράς και παρόλα αυτά ε, διαπραγματεύεται. Δηλαδή ε, σκεμμένα και γνώση της παραβίαση του νόμου. Τι γίνεται με τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τι συμφωνία είναι αυτή και θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν είναι ε, ευθυγραμμισμένη με το GDPR αυτή η συμφωνία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νομίζω δεν είναι σωστή εδώ στη στάση της. Λέει είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Και τι θα γίνει μετά με την Κίνα, με τη Βραζιλία, με την ε, Ρωσία και πού τελειώνει αυτή η ιστορία. Αν δεχτούμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα υπαγορεύουν διμερείς συμφωνίες με κράτη-μέλη, με την Κίνα τι θα κάνουμε, γιατί γίνεται και προηγούμενο εδώ. Τα μέλη του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ε, ε, εάν δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για μια διευθυντή συμφωνία, θα παραμείνει στον αιώνα τον άπαντα, γιατί δεν έχουμε την εξουσία να την αναστείλουμε, να την ανακαλέσουμε. Να είστε λοιπόν πάρα πολύ σίγουροι ότι όταν ψηφίζετε μια συμφωνία είναι πραγματικά κλειδωμένη ε, νομικά. Καλά, ε, υπάρχει το έμλας, υπάρχει εργαλείο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ως συνήθως, τη γνωστή της τακτική. Ε, το δοκιμάσαμε είναι αργό. Μα δεν το έχουμε δοκιμάσει καν. Δεν έχει γίνει καμιά σοβαρή απόπειρα να βελτιωθεί. Και βεβαίως, στο ένα κράτος δημοκρατικό, κράτος δικαίου, καμιά φορά οι διαδικασίε αργούν. Ε, στις δικτατορίες είναι συνοπτικέ και δαχείε οι διαδικασίε. Εμείς ε, έχουμε πάρα πολύ καλού λόγους για να υπάρχει δικαστικό έλεγχο και δεν μπορούμε να το καταργήσουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Ε, πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται. Ναι. Το Ρινιού πήρε το λόγο. Θα πάρετε κι εσείς το λόγο, αλλά να συνεχίσουμε τις πολιτικές ομάδες. Και μετά θα δώσουμε το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Πράσινο δεν βλέπω. Παρόντα. Α, βλέπω. Ο κύριος Μπράιερ. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ θετικό που έχουμε εδώ τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων ε, και που ε, γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την συμμόρφωση ε, του Ευρωπαϊκού Νομικού Συστήματος σε αιτήματα από άλλες χώρες για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή και μεταδεδομένων. Επομένως, ε, χαιρετίζω πραγματικά τα όσα ακούσαμε. Θα πρέπει να θυμηθούμε τα εξής. Δεν έχουν πραγματική προστασία ε, για την ε, βάση, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ούτε για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, μια και τα συζητάμε και τα αναφέρουμε εδώ. Επίσης, δεν υπάρχει ανεξάρτητη αντιμετώπιση όσον αφορά τον χειρισμό των δεδομένων και μερικές φορές δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική εκ των ε, αποκατάσταση ε, και επομένως ε, δεν είναι δυνατόν τέτοιου είδους προσωπικά στοιχεία τα οποία καλύπτονται από το GDPR να μεταφέρονται στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Θέλουμε πραγματικά να ενδυναμώσουμε και να κυρώσουμε, να τιμωρήσουμε την μεταφορά δεδομένων, γιατί χωρίς τιμωρία δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Εάν τιμωρήσουμε, αν υπεβάλλουμε κυρώσεις σε ε, ε, εταιρείε ε, οι οποίες παραβιάζουν τον νόμο, τότε θα έχουμε χάσει τον, τη μάχη αυτή απέναντι στις ΗΠΑ. Δεύτερη ερώτηση, βλέποντας και διαβάζοντας αυτήν την Cloud Act, θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πάροχοι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένε Πολιτείε, μια και ε, θα έχουν την δυνατότητα να μεταδίδουν, να μεταφέρουν ε, παράνομα ε, στοιχεία τέτοιου είδους στις Αμερικανικές αρχές. Επίσης, το αίτημα για νομική αδειοδότηση, ας πούμε, ε, σε ποιες περιπτώσεις ε, θα δίνεται σε, Thank you. Ε, σε ποιες περιπτώσεις θα δίνονται οι άδειε έτσι ώστε να μεταφέρονται τα στοιχεία αυτά στα δικαστήρια. επόμενη ομιλήτρια, κυρία Κάνκο. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι σιγά σιγά θέλουμε να ε, ε, να ξεφτύσει η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, εδώ θα πρέπει να δούμε το θέμα όχι μονάχα σε σχέση με την Αμερική αλλά και σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Είναι γενικώ ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειαζόμαστε συνεργασία σε διεθνές επίπεδο επί πολλών θεμάτων. Ε, η Ιαπωνία ας πούμε είπε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς ε, ε, διεθνή πρότυπα και διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας. Ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξής. Η Κομισιόν και η Επιτροπή θεωρεί ότι ε, πρέπει να αλλάξουν οι συμφωνίες σχετικά με την ροή ε, δεδομένων μεταξύ των G7 και των G20. Επίσης, ε, η τροποποίηση των προτύπων προστασίας είναι δυνατή υπό την παρούσα διοίκηση. Επίσης, σε σχέση με τις χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός του πεδίου, εάν ας πούμε έχουμε μία χώρα λιγότερο αναπτυγμένη όσον αφορά την προστασία των δεδομένων κτλ. Τι θα κάνουμε ε, σε τέτοιες ε, περιπτώσεις, γιατί εδώ έχουμε στοιχεία τα οποία αποτελούν διεθνείς προκλήσεις. Η κυρία Ντάλη, ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως αυτά είναι πολύ γενικά ζητήματα. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ε, ότι είναι απόλυτο, ε, ε, δεν κάνουμε μια συζήτηση χωρίς την Κομισιόν. θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. γιατί ενδεχομένως ας πούμε θα μας πει ότι θα πρέπει σε ποινικέ περιπτώσεις να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αδίκημα και πώς περιγράφονται τα αδικήματα, γιατί στα διάφορα νομικά συστήματα η περιγραφή δεν είναι και ο ορισμός δεν είναι ίδια. Επίσης υπάρχουν ας πούμε η Google, η Facebook, η Twitter ε, που ε, θα πρέπει να δούμε πώς προστατεύουν και αν προστατεύουν τους χρήστες τους ε, ε, όσον αφορά την προστασία των προσωπικών των ε, δικαιωμένων. Επίσης, όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την προστασία προσωπικών δεδομένων, ξέρουμε ότι έχει υπογραμμιστεί ότι οι διεθνείς συμφωνίες μπορεί να εφαρμοστούν, αλλά μονάχα εάν η άλλη ετούμενη χώρα παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα δύο σημεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Το ζήτημα είναι πώς θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στις 11 προϋποθέσεις ε, του EDPS. Ε, Αυτό είναι το θέμα, γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Ε, η ίδια η δικιά μας νομική υπηρεσία δεν ε, έδωσε συγκεκριμένη απάντηση. Ε, θέλω να πω ότι στην γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας δεν είδαμε ισχυρή επιχειρηματολογία όσον αφορά αυτά τα θέματα, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία είναι να λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και θα σέβεται και τις διατάξεις του του GDPR, αλλά παρόλα αυτά εδώ νομίζω ότι έχουμε ένα τετραγωνισμό του κύκλου που δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστούμε για όλο σας το έργο. Ναι σαφή τα συμπράσματα. Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βρεθούν ε, μεταξύ κάποιες αντιφατικής νομοθεσίας ε, που θα προκύπτει από το US Cloud και το GDPR. Και για να έχουμε ασφαλεία δικαίου είναι σημαντικό να συνάψουμε μία συμφωνία ε, που θα εξαλείφει αυτές τις συγκρούσεις. Θα πρέπει αυτή η συμφωνία επίσης να υπερισχύει υπέρ του από το δευτερογενές δίκαιο της Ένωσης κάλεσε και την Κομισιόν συνάδελφο Ντάλι, Μα είπαν ότι είναι εδώ. Έτσι λοιπόν το δικό μα μήνυμα προ την Κομισιόν πρέπει να είναι σαφέ. Εμεί. δεν θα συνενέσουμε ω Κοινοβούλιο σε οποιαδήποτε συμφωνία που δεν θα σέβεται ε, τα πρότυπα τη δευτερουργής νομοθεσία και δεν θα έχει ισχυρέ ασφαλιστικέ δικλείδε για το διτό αξιόπινο, πλήρη αμοιβαιότητα ε, και ε, ισχυρά δικονομικέ και μάλλον ισχυρέ δικλείδε για τα δικονομικά δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και το μήνυμα στο Συμβούλιο πρέπει να είναι σαφέ. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα επίπεδα προστασία για όλου του Ευρωπαίου πολίτε και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να μπουν σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι γι' αυτό. Ως Ευρωπαϊκή Συμφωνία θα πρέπει να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Συμφωνία θα πρέπει να έχει πολύ ισχυρές δικλείδες και θα πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Σας ευχαριστώ. Σας ακούσουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρότεινα να πάρετε το λόγο για μια σύντομη παρέμβαση. Γιατί έγιναν διάφορες αναφορές στο ρόλο της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που υλοποιούνται από το Συμβούλιο. Ας ακούσουμε την κυρία Ντεφρεπού, πιστεύω. Εκπροσωπείτε την Κομισιόν εδώ. Και επιμένω έχουμε και ένα επόμενο σημείο που θα σας δώσω λεπτά και έχουμε και ακόλουθη συζήτηση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ γιατί στις 11.30 ε, θα έρθουν και οι βουλευτέ από την ΕΚΟΝ. Παρακαλώ, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Λέγομαι Ιζαμπέλ Περινιόν ε, και είμαι ε, αρμόδια για ποινικέ υποθέσει. Ακούσαμε τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου και θέλω να κάνω τρία σχόλια και κατόπιν θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο που είναι αρμοδίο για την προστασία των δεδομένων. Για το πρώτο σημείο. Εμείς διαπραγματευόμαστε βάσει εντολή που λαμβάνουμε και στην εντολή αυτή, αυτή η εντολή μάλλον είναι σαφής και θέλουμε να έχουμε ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δεδομένων και τα θεμελιώδη δικαιώματα και δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Επίσης έχουμε δεσμευτεί και ήταν σαφές ε, ιδίως κατά την ακρόαση Επιτρόπου Ρέντερς ότι δεν θα υπογράψουμε καμία συμφωνία πριν να έχουμε μία συμφωνία μαζί σας μετά τους τριμερεί διαλόγους για τους εσωτερικούς κανόνες ε, πριν να υπογραψούμε οτιδήποτε με τους Αμερικανούς. Και το μήνυμα που επαναλαμβάνουμε σε αυτούς είναι αυτό. Δεύτερον, για τη συμφωνία, με, για τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ηνωμένο Βασίλειο, είπα. Έχουμε στείλει πολλές επιστολές και τους εξηγούμε ότι έχουμε ανησυχίες. Και αφού υπεγράφει συμφωνία, επίσης στείλαμε σαφέστατη επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξηγήσαμε ότι έχουμε ανησυχίες επί της συμφωνίας και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο είναι σαφέστατο και το διευκρινίσαμε και στους Αμερικανούς ότι η συμφωνία που έχουν υπογράψει με τους Βρετανούς δεν είναι το μοντέλο που θέλουμε να ακολουθήσουμε και ζητήσαμε εξηγήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μας ανησυχούν. Τρίτο σημείο. Για την ε, αμοιβαία νομική συνδρομή και την ε, σχετική σύμβαση που έχουμε με τη ΣΥΠΑ. Εμείς ε, θέλουμε συνεχώς να βελτιώνουμε την ΕΜΛΑΤ και είχαμε συζητήσεις με τους Αμερικανούς, ε, συνεχίζουμε τις πιέσεις ε, και έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την ΕΜΛΑΤ. Αλλά δυστυχώς δεν αρκεί αυτό. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο και να συνέψουμε μια άλλη συμφωνία με τις ΗΠΑ, γιατί ξέρουμε ότι θα πρέπει να θέσουμε τέλος σε μια πρακτική που δεν μας δίνει αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες. Τώρα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο για την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετείχαν στη συζήτηση από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία των Δεδομένων και την Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου τόνισαν όλοι τη σημασία του να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που έχουμε στον τομέα της επιβολής του νόμου. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει η ΕΜΛΑΤ αυτά σε όλες τις περιπτώσεις. Και όλοι εξέφρασαν υποστήριξη ως προς να ε, βρούμε ένα μέσο που να επιτρέπει άμεσα αιτήματα και καλώς όρισα και τη συμφωνία. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε μια διεθνή συμφωνία έτσι ώστε να ρυθμίζεται το πώς μπορούμε να ελοποιούμε τα άμεσα αιτήματα. Παρά να έχουμε παραδείγματος χάρη άμεσα αιτήματα δυνάμει του Cloud Act και μπορεί να οδηγήσει αυτό σε συγκρούσεις νομοθεσίας και οι πολίτες μπορεί να μην λάβουν την προστασία που χρειάζονται και θα μπορούσαμε να έχουμε πιθανόν ε, μια κατάσταση σύγκρουσης νομοθεσίας. Έτσι λοιπόν ε, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση σύγκρουσης των νομοθεσιών διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Φυσικά υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων, αλλά και δικονομικέ ε, ασφαλιστικές δικλείδες. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η συμφωνία, αν τη συνάψουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, θα περιδοτούσε μια συμφωνία ομπρέλα. Η, η Συμφωνία Προστασίας των Δεδομένων που τέθηκε σε ισχύ νομίζω το Φεβρουάριο του 2017 με μεγάλη υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δίνει ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας των δεδομένων. Είναι εφαρμοστέα αλλά χρειάζεται να υπάρξει και μία συμφωνία μεταφορά, μία συμφωνία διαβίβασης. Και αυτή τη συμφωνία θα διαπραγματευτούμε και θέλουμε να συνάψουμε τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή είναι θετικό να έχουμε μία τέτοια συμφωνία γιατί ουσιαστικά σχετίζεται με τη συμφωνία Ομπρέλα. Αν έχετε δει την εντολή που λάβαμε από το Συμβούλιο έχει ως στόχο να προσαρμόσει τη Συμφωνία Ομπρέλα στη συγκεκριμένη περίπτωση της άμεσης συνεργασίας. Έτσι λοιπόν πάμε ε, περαιτέρω και θέλουμε να προσαρμόσουμε αυτή τη Συμφωνία Ομπρέλα για να την προσαρμόσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Φυσικά, ακούμε πολύ σοβαρά όλες τις ανησυχίες και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε με τη ΣΥΠΑ ότι έχουμε μια συμφωνία προστασίας. Και δύο λόγια ακόμη γι' αυτό. Όλοι θα πρέπει να έχουμε κατά νου και άλλες συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο Στρασβούργο με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, για την σύμβαση της Βουδαπέστης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Πρόκειται για μια πολυμερή συμφωνία όπου συμμετέχουν 64 κράτη, μέρη και έχει ευρύτερο πεδίο έτσι λοιπόν έχουμε διάφορα μέσα εδώ σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία στο θέμα της επιβολής του νόμου. Και φυσικά θα προσπαθήσουμε να δυσφαλίσουμε τις απαραίτητες δικλείδες. Λοιπόν, κινδυνεύουμε να καθυστερήσουμε χρονικά. Είδα ότι η κυρία Ιντβελτ ήθελε να δώσει μια σύντομη απάντηση. Να είστε σύντομοι παρακαλώ έτσι ώστε να έχουν και χρόνο οι ομιλητές να απαντήσουν. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η Κομισιόν μας είπε ότι λαμβάνει σοβαρά όλες τις ανησυχίες. Ε, από ό,τι φαίνεται όχι και τόσο. Διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να περιμένετε να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις μέχρι να έχει υιοθετηθεί το θέμα για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Θα πρέπει μετά να ξεκινήσετε τις διαπραγματεύσεις, γιατί αυτό μας είχε υποσχεθεί η Κομισιόν, να γνωρίσετε εντελώς ε, τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Πόπτη. γιατί Δεύτερον, η ΛΥΜΠΕ μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία πλήρη γραπτή έκθεση για όλα όσα έχουν γίνει για να βελτιωθούν οι έμλα ε, οι συνθήκες αμοιβαζομικής συνδρομής και γιατί απέτυχαν, γιατί μία προφορική δήλωση δεν μας αρκεί. Τέλος, είπατε ότι έχετε ανησυχίες για τη συμφωνία είπα Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι απλό, είτε σέβεται το GDPR είτε όχι. Αν το σέβεται, πολύ ωραία. Αν όχι, τότε δεν θα πρέπει να ανησυχείτε, θα πρέπει να ξεκινήσετε διαδικασία επί παραβάση. Σημειώνουμε το έτοιμά σας. Θα διαβεβαιστεί αρμοδίως στου συντονιστάς για να ληφθεί η απόφαση και να στείλει ε, επιστολή ο Πρόεδρος στην Επιτροπή. πέντε λεπτά ο καθένας για να απαντήσετε τώρα, τα μέλη του πάνελ μας. Ε, από το επόπτη προστασία προσωπικών δεδομένων, ο κύριος Βιβορόφσκι. Για λόγους χρονικού θα απαντήσω μόνο κάποια από τα ερωτήματα που ακούσαμε. Βεβαίως θα σας ε, απαντήσουμε εκτενέστερα. Ε, και μόνο το γεγονός ότι πρώτα προτείνουμε ε, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ακριβώς αυτό κατατείνουν, ότι χρειάζεται να λυθεί αυτό το θέμα πριν αποφασίσουμε τι κάνουμε με τις τρίτες χώρες. Για μας ήταν προφανές, γι' αυτό κάναμε και αυτή την παρουσίαση. Ελπίζω να ε, σημειωθεί σύντομα πρόοδος εκεί, μαζί με τη συζήτηση για τη γενικότερη συμφωνία ε, ομπρέλα, όπως λέγεται. Επίσης χαίρομαι πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε προς το παρόν προφορικά μόνο για τις βελτιώσεις που προτείνουν για το ΕΜΛΑΤΣ Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Τώρα βρίσκομαι στην εξή δινή κατάσταση. Δεν μπορώ να εκτιμήσω τη συμφωνία είπα, Ηνωμένου Βασιλείου που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο γιατί δεν εμπίπτει στη δική μας ε, δικαιοδοσία αυτό. Ο Ευρωπαίος Υπόπτης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ασχολείται με τις διμερείς συμφωνίες. Άρα θα ζητήσουμε να μας ενημερώσει η ε, ομόλογός μας του Ηνωμένου Βασιλείου ε, για το πώς μεταφράζονται όλα αυτά στην πράξη και τι σημαίνουν και αν περιλήφθηκε στις διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς μιας ενδεχόμενης συμφωνίας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. μιλώ για την Αμερικανική πλευρά. Θα είναι διεθνή συνθήκη ή εκτελεστική συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Το θυμόμαστε από παλαιότερες συμφωνίες ε, στις εμπορικές συμφωνίες ας πούμε ε, που συμφωνούνται από ε, οι πολιτείες μεμονωμένες ή από το ομοσπονδιακό επίπεδο. Το συγκεκριμένο δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδος συμφωνίας είναι. Ε, σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες λύσεις, που θα μπορούσαμε επίσης να λάβουμε υπόψη και ιδιαίτερα το ρόλο ε, τη Σύμβαση για το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ε, μπορεί ε, να ε, είναι μια ακαδημαϊκή ανησυχία. Αν δούμε στο χάρτη ποια είναι τα μέλη εκεί, υπάρχουν δύο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ε, συμβληθεί και μία χώρα από αυτές είναι η Ιρλανδία. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει πολύ ε, την υλοποίηση της συμφωνίας. Δεύτερον, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν και Τουρκία είναι συμβαλόμενα μέρη, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό, και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ιαπωνία δεν είναι οι μόνες χώρες για τις οποίες συζητούμε ε, όταν πρόκειται για πρακτική ανταλλαγή δεδομένων. Θυμάμαι τις εποχές που υπογράφηκε αυτή η συμφωνία από το 99 με το 2001 και η συζήτηση ήταν επί της ουσίας και όχι επί της διαδικασίας τότε. Παραμένουμε ε, είμαστε στη διάθεσή σας προσέχουμε αυτά τα θέματα και τα παρακολουθούμε ε, ευχαριστώ κύριος Μπεν ε, ευχαριστώ πρόεδρε Θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά νομίζω ότι ε, ήδη απαντήθηκαν. Υπήρχε και μία ερώτηση από την κυρία Ζήπελ, αν δεν κάνω λάθος, ε, σχετικά με τι σχέσει ανάμεσα στη συμφωνία ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο και το Privacy Shield πώς να σας το πω. Μέχρι τώρα το Privacy Shield και το Cloud Act ήταν κατά κάποιο τρόπο δύο χωριστά πράγματα. Ωστόσο έχετε δίκιο, ε, είναι πολύ ουσιαστική η ερώτησή σας. Ένας από τους λόγους που ήταν ξεχωριστά ε, τα δύο στοιχεία ήταν γιατί δεν υπήρχε συμφωνία. Τώρα υπάρχει μια διμερής συμφωνία όντως, όντως ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει κάποιο αντίκτυπο και θα το δούμε, θα το ελέγξουμε ε, στα πλαίσια του Privacy Shield. Θα δούμε δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία, όταν θα έχουμε και όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας, πώς εμπλέκονται τα, τα μεν με τα δε. Ε, όσον αφορά τα όσα ρώτησε ο κύριος Πράιερ, όντως εδώ έχουμε μία πρώτη αξιολόγηση μονάχα. Είναι ε, πρώτη αξιολόγηση καθότι δεν έχουν υπάρξει ακόμα καταγγελίες όσον αφορά το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιος όμως ότι ε, θα υπάρξουν ε, τέτοιες καταγγελίες και εάν αυτή είναι η τελική μας θέση, οπωσδήποτε θα πρέπει να ενδυναμωθεί γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Επίσης, σε σχέση με την χρήση των υπηρεσιών ε, του νέφους Cloud Services, ε, πρέπει να δούμε ε, ποιες είναι οι διαρθρώσεις που μπορούν να υπάρξουν σε σχέση με το άρθρο 28 του GDPR Τώρα, σύμφωνα με αυτά που έχω γράψει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων. Εάν λησμόνησα κάτι, παρακαλώ να μου το θυμίσετε. Monsieur Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω ομαδοποιημένα να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, ε, πρώτα απ' όλα το θέμα των συγκεκριμένων μέτρων ε, που ανέφερε η κυρία Ζήπελ όσον αφορά την, τις συμβάσεις δικαστικής συνδρομής στα ΕΜΛΑΤΣ. Ε, υπάρχει, υπάρχουν στο πρωτόκολλο για, την, κυβερνο, για το κυβερνοέγκλημα πορά στοιχεία τα οποία μπορούν να αναφερθούν σε αυτόν επίσης υπάρχουν και οι έκτακτες και ε, συνοπτικές ε, διαδικασίες. Ε, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει τις, τη νέα γενιά των ΕΜΛΑΤΣ και βεβαίως εάν θέλουμε να προχωρήσουν και τα κνήλστα θα πρέπει να δούμε και τις διαδικασίες οι οποίες υφίστανται ήδη αλλά και να δούμε και ποια είναι τα μέσα τα οποία ενδεχομένως θα έχουμε έτσι ώστε να λειτουργήσουν σωστά τα εργαλεία που θα θα έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, ε, το Κομιτέ Ευρωπαίο υπενθύμησε ότι ρόλος του είναι να ελέγχει τη συμμόρφωση της αποκάλυψης ε, σύμφωνα με τους ε, ε, σύμφωνα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ότι η αποκάλυψη θα πρέπει να γίνεται ε, υπό την επιτήρηση των Ευρωπαϊκών Αρχών. Ε, να μην το ξεχνούμε αυτό. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπε και ο Κάρστεν προηγουμένως, ε, στην κατάσταση που περιέγραψε προηγουμένως, ε, η εγγύηση του Privacy Shield δεν εφαρμόζεται αλλά ε, σε παράρτημα της επιστολής που μας απευθύνεται, διαφαίνεται η πρόθεση τουλάχιστον να ληφθούν υπόψη οι επόμενες εκτελεστικές αποφάσεις που θα, ε, συνάψει ε, θα συνάψουν οι ΗΠΑ Πολιτείες με άλλες χώρες, όχι απαραίτητα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, το ανέφεραν αυτό οι δύο προλαλήσαντες, εμείς δεν έχουμε δικαιοδοσία να ελέγξουμε το κατά πόσον έχουν δικαίωμα οι χώρες ή ε, αρμοδιότητα ε, να προχωρούν σε τέτοιες συμφωνίες. Το θέμα είναι να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εάν προχωρήσουμε στην οδό των διμερών συμφωνιών με τις διάφορες χώρες, ε, θα υπάρξουν οπωσδήποτε διαφορές όσον αφορά τις διαδικαστικές ε, εγγυήσεις από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να ε, δούμε κατά πόσον οι δικονομικές διατάξεις και εγγυήσεις διαφέρουν πολύ μεταξύ των χωρών, έτσι ώστε να έχουμε μια ιδέα του πόσο μπορεί να διαφέρουν και οι εγγυήσεις στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ναι, έχουν τεθεί κάποιες ανησυχίες και είναι σαφές ότι είναι βάσιμες. Περιγράφεται μια κατάσταση που παραμένει ανοιχτή, καθώς είναι ανοιχτή και η διαδικασία. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και υπάρχει η προοπτική σύνεψη συμφωνίας με τις ΗΠΑ που μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επαρκείς εγγύσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που προστατεύονται από τη χάρτα των Ευρωπαϊκών των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο άρθρο 8 για την ιδιωτικότητα. Είναι μια κατάσταση λοιπόν που μας ανησυχεί, πρέπει να την παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και αυτό θα κάνουμε. Είναι ανοιχτή λοιπόν η κατάσταση. Το επόμενο σημείο επίσης αφορά την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια άλλη έκθεση που θα ακούσουμε για ένα άλλο θέμα που μας ανησυχεί, που είναι το δικαίωμα στη διαγραφή δεδομένων που έχουν αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα που προστατεύονται από τη χάρτα. Πρόκειται για ένα σημείο που αφορά την προστασία των δεδομένων, τις ιστοσελίδες και την εφαρμογή της οδηγίας που αφορά την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης να διασφαλίσει τα δεδομένα και να προστατεύσει τα δικαιώματα. Όμως, παρατέταρτο, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν θα έλεγα να αποχαιρετήσουμε τους ομιλητές μας και να ετοιμαστούμε για το επόμενο σημείο. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμη, κυρία Ζήπελ, ίσως απλώς για να καλύψω το χρόνο μέχρι το επόμενο σημείο. Γιατί η σημερινή συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής, ε, με ανησύχησε κάπως. Με ανησύχησαν αυτά που ακούσαμε. Και ακόμη και αν συμφωνώ με την ιδέα της κυρίας Σίντεβελτ για την επιστολή, νομίζω, νομίζω ότι θα πρέπει να διευρυνθεί. Γιατί τι βλέπω επίσης, ότι προφανώς η Κομισιόν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη ε, τις ε, αρμοδιότητες και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας ε, λένε ότι το e-evidence αποτελεί νομική βάση για μια διεθνή συμφωνία και από την άλλη έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Αναρωτιέμαι σε ποια βάση δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα για τις ε, ηλεκτρονικές αποδείξεις, αλλά για τι πράγμα μιλάμε. Και τελικά προσπαθούν να προκρίνουν ε, το αποτέλεσμα της νομοθεσίας της ηλεκτρονικής αποδείξης στις διαπραγματεύσεις τους. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε λοιπόν και άλλες ερωτήσεις πρέπει να θέσουμε πέρα από αυτές που μας είπε η Σόφη και θα πρέπει να κάνουμε σοβαρότερε συζητήσει για τους φακέλους αυτούς. Κύριε Μπράιερ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση έθεσα στην νομική υπηρεσία. Μπορώ να ζητήσω να μου απαντήσουν για το τι σημαίνει η δικαστική έγκριση και τι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή έννοια αυτή. Θέλετε να σχολιάσετε παρακαλώ νομική υπηρεσία. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Συγγνώμη. Δεν δούλευε. Λοιπόν, για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να το δούμε ένα περίπτωση, αλλά υπάρχει νομολογία του δικαστηρίου για το τι πρέπει να εννοούμε ως δικαιοδοσία. Υπάρχουν κριτήρια. Πρόκειται για ένα δεδομένο όργανο που ουσιαστικά είναι αμερόληπτο απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Είναι ανεξάρτητο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, ανάλογα με τα όργανα που στοχεύονται, αν μπορεί να θεωρηθούν ή όχι δικαιοδοσίε. Σχόλιο εκτό μικροφώνου, τον κύριο Μπρέιερ. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα να σας απαντήσω στην ερώτηση αυτή. Αν ε, θέλουμε να ξέρουμε αν ε, είναι δικαιοδοτικό όργανο ένα όργανο στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να δούμε αν είναι ανεξάρτητο το όργανο αυτό για να θεωρηθεί δικαιοδοτικό. Ίσως για να απαντήσω και στις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις της κυρία Σίπελ. Διακοπή του μικροφόνου σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της αρμαδιότητας του κράτους μέλους να διαπραγματευτεί δική του συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο βαθμό που δεν έχει ασκήσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά αφού θα έχει συμφωνηθεί μια νέα συμφωνία, μετά το κράτος μέλος ε, δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα κανονικά και για το θέμα της διαδικασίας ε, της κύρωσης της συμφωνίας αυτής και το ρόλο του Αμερικανικού Κογκρέσου, είναι σαφές ότι το Cloud Act, για το Cloud Act ε, χρειαζόμαστε έγκριση από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Τώρα Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και άλλη μια παρουσίαση από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δικαίωμα που αφορά το δικαίωμα στη λύθη και τη διαγραφή των δεδομένων. Σε ένα λεπτό. Oh. As said, got some 45 minutes. Έχουμε 45 λεπτά προγραμματίσει για το εξή θέμα στην ημερήσια διαταξή πριν την κοινή μα συζήτηση με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Είναι τα σημεία 14 και 15, παρουσίαση των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της 24 η Σεπτεμβρίου, στην υπόθεση 136 κάθετος 17 σχετικά με την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες. Και το 15 αφορά μια άλλη υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης. Είναι το λεγόμενο δικαίωμα στη λύθη ένα πρόσωπο έχει το δικαίωμα τα προσωπικά του δεδομένα ε, ε, να αφαιρούνται ε, όταν έχουν τύχει αθέμητης ή παράνομης επεξεργασίας. Mrs. Olga Έχουμε την κυρία Όλγα Χστρόβα. Τι όνομα είναι αυτό. Δύσκολο να το προφέρω. Το συγγνώμη. was a great pronunciation. Πολύ ωραία το είπατε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή και το λόγο που μου δίνετε. Μας ζητήθηκε να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή σας τις δύο αποφάσεις που είναι και οι δύο της 24ης Ενάτου του 2019. Οι δύο αυτές ε, ε, αποφάσεις είναι η ε, απάντηση σε προδικαστικό ερώτημα ε, από το Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας και τα δύο για την ερμηνεία της τότε οδηγίας για την προστασία των προσώπων ε, στην ε, εξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο μεταξύ έχει αντικατασταθεί η οδηγία αυτή από το GDPR, αλλά το δικαστήριο εξέτασε και τα δύο πεδία εφαρμογής και της οδηγίας και του κανονισμού και εξέδωσε απόφαση και απάντηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα πλαίσια του GDPR στο μέλλον. Ανέφερε ο πρόεδρος ε, αυτά τα δύο και βασίζονται και στην απόφαση Google κατά Ισπανίας του Μαΐου 2014. Θυμίζω για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημερινή απόφαση το εξής. Στην υπόθεση Google κατά Ισπανίας ε, το δικαστήριο ε, έθεσε το δικαίωμα στη λύθη, στο δικαίωμα της αφαίρεσης ε, προσωπικών δεδομένων και είπε το δικαστήριο ότι οι ε, πολίτες, τα ε, πρόσωπα έχουν το δικαίωμα στη λύθη και μπορούν οι σελίς, οφείλουν μάλλον να αφαιρούν το περιεχόμενο όταν υπάρχει λόγος, τη διαγραφή των συνδέσμων ε, που μπορεί κανείς να βρει στοιχεία βάζοντας σε μια μηχανή αναζήτηση το όνομα του προσώπου. Ε, η σημερινή απόφαση ε, διευκρίνησε σημαντικά το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της διαγραφής των συνδέσμων και οι μηχανές αναζήτησης τύπου Google θα πρέπει να το σέβεται αυτό όταν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Θα επικεντρωθώ πρώτα στην υπόθεση Google C507 κάθετος 17. Είναι το δικό σας θέμα 15, το δεύτερο από τα δύο. Και έχει να κάνει με τα γεωγραφικά ε, όρια του δικαιώματος στη διαγραφή ε, συνδέσμων. Αυτό προέκυψε από μία διένεξη που είχε Google με την ε, γαλλική ΚΝΙΛ ε, η οποία είχε ζητήσει να ε, κάνει η Google διαγραφή συνδέσμων σε όλες τις επεκτάσεις ε, αναζήτησης του πεδίου, δηλαδή παγκόσμια. Αρνήθηκε η Google να το κάνει και έβγαλε τους συνδέσμους μόνο από την έρευνα που γίνεται σε το name, name από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό ε, κατέληξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ε, η Google έκανε έφεση απέναντι σε ένα πρόστιμο που της επέβαλε η CNIL. Στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προδικαστικό ερώτημα το Συμβούλιο της Επικρατείας Γαλλίας και ρωτούσε ακριβώς αν θα πρέπει αυτό να γίνει παγκοσμίω στι μηχανές αναζήτησης ή μόνο στη μηχανή αναζήτησης που αντιστοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα domain ε, names ή ακόμα και σε εκείνα που αντιστοιχούν σε κράτη-μέλη ε, που ζητήθηκε η διαγραφή των συνδέσμων. Στη συνέχεια, επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ε, το Γαλλικό, ρώτησε τι τεχνικές γεωγραφικού αποκλεισμού χρησιμοποιεί η Google και αν αυτό ισχύει και αναφερόμαστε και στην απόφαση ε, της ε, ε, Google κατά Ισπανίας. Στο άρθρο 17 του GDPR καλύπτεται η διαγραφή συνδέσμων τώρα. Είναι το δικαίωμα στη διαγραφή και στο δικαίωμα στη λύθη. Η αναφορά αυτή. Για να ξεκαθαριστεί το εδαφικό πεδίο της διαγραφής συνδέσμων, θύμισε πρώτα το δικαστήριο το στόχο του GDPR και της προηγούμενης οδηγίας ε, δηλαδή να υπάρχει εγγυημένο υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Από τη μια λοιπόν το, το δικαστήριο δέχτηκε ότι η παγκόσμια διαγραφή συνδέσμων ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτό το στόχο. Το ε, ίντερνετ δεν γνωρίζει σύνορα. Μια τέτοια μηχανική αναζήτηση, μηχανή αναζήτηση, συγγνώμη, έχει πληροφορίες παντού και, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Σύμφωνα με το δικαστήριο, αυτό δικαιολογεί την ύπαρξη δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσει από μια μηχανή αναζήτηση να κάνει διαγραφή συνδέσμων παγκοσμίω. Από την άλλη, συνεχίζει το δικαστήριο και τονίζει ότι πολλέ τρίτε χώρε δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα διαγραφή συνδέσμων ή έχουν άλλη ερμηνεία και άλλη προσέγγιση στο δικαίωμα αυτό. Και το δικαίωμα προστασία προσωπικών δεδομένων δεν είναι απόλυτο. Θα πρέπει να το βλέπουμε σχετικά ε, με τη λειτουργία του στην κοινωνία και ε, σε αντιστάθμισμα άλλων ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή η στάθμιση βεβαίως διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα, ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια το δικαστήριο ε, αναφέρει ε, το GDPR και την οδηγία. Ιδιαίτερα το άρθρο 17 του GDPR, παράγραφος 3 μικρό α, ε, ε, ο Ευρωπαίος νομοθέτης ε, βρίσκει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων από τη μια και την προστασία της ιδιωτικότητας και από την άλλη ε, στο δικαίωμα στην πληροφορία και την ελευθερία των χρηστών του ίντερνετ. Και αυτό το πράττει μόνο στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προκύπτει από καμία διάταξη ούτε της οδηγίας ούτε του κανονισμού ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης θα ε, είχε ένα πεδίο εφαρμογής που θα υπερεύαινε ε, την επικράτεια των κρατών μελών. Συμπεραίνει το Συμβούλιο ότι δεν υπάρχει υποχρέωση βάσει ευρωπαϊκού δικαίου η διαγραφή συνδέσμων να γίνεται παγκοσμίω. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση αν η διαγραφή συνδέσμων θα πρέπει να γίνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο σε ένα κράτος μέλος, το, Δικαστήριο θύμισε ότι ο Ευρωπαίος νομοθέτης επέλεξε τη μορφή του κανονισμού ως νομικού μέσου ακριβώς για να υπάρχει παντού υψηλού επίπεδου συνεπής εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η διαγραφή συνδέσμων καταρχήν θα πρέπει να γίνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα λέει το δικαστήριο ότι ε, και μάλιστα βάσει βάση το άρθρο 85 του GDPR διαφέρει η αίσθηση ενημέρωσης από χώρα σε χώρα ε, και δικαιώματος ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων με το δικαίωμα στην ενημέρωση και την ελευθερία έκφραση. Για το γεωγραφικό προκλεισμό ήταν σύντομο το δικαστήριο και είπε ότι η μηχανή αναζήτηση θα πρέπει να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία του ενδιαφερμένου προσώπου, τα οποία είτε θα προλαμβάνουν ή τουλάχιστον θα αποθαρρύνουν σοβαρά χρήστες του διαδικτύου στα κράτη-μέλη να προσφεύγουν σε συνδέσμους που ε, υπόκεινται στη διαγραφή. Σύντομα, αν θέλετε να συνοψίσω πιο πρακτικά την απόφαση του δικαστηρίου, βασικά λέει ότι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση της μηχανικής αναζήτησης μηχανή αναζήτηση να κάνει διαγραφή συνδέσμων παγκοσμίω. Δηλαδή, ο πάροχος θα πρέπει να αφαιρεί ε, κάποιους συνδέσμους ε, ως αποτελέσματα αναζήτησης μόνο στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Ωστόσο, ε, δεν απαγορεύεται τέτοια πρακτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προβλέπονται εξαιρέσει και η αρμόδια εθνική αρχή κάθε φορά θα πρέπει να σταθμίζει τα δικαιώματα που διακυβεύονται με βάση τα εθνικά πρότυπα και να ε, ζητεί από τη μηχανή αναζήτησης να τα φέρει από όλη την επικράτειά του. υπάρχουν μέτρα που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τον γεωγραφικό αποκλεισμό για να μην έχουν πρόσβαση χρήστες ε, εκτός Ένωσης. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη απόφαση η οποία καθόρισε το, μάλλον διευκρίνησε ε, το ρόλο ε, των ε, φορέων εκμετάλλευσης. Είναι η υπόθεση 136 κάθετος 17. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα ζήτησαν από την Google να διαγράψει συνδέσμους που είχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως πολιτικές απόψεις, θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Ε, και στις τέσσερις περιπτώσεις η Google απέρριψε το αίτημα, οπότε ε, πήγαν στην ΚΝΙΛ οι ε, ετούντες και τελικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας στη Γαλλία. Θα ήθελε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας να γνωρίζει εάν η απαγόρευση για ειδικέ κατηγορίες δεδομένων αφορά και τη μηχανή αναζήτησης. Δηλαδή, η Google θα πρέπει να συμμορφωθεί ε, με τις διατάξεις ε, και την επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης, ζήτησε μια διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογή και την επεξεργασία δεδομένων σε ό,τι αφορά ε, καταδίκες, ποινικέ και αδικήματα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, θύμισε το δικαστήριο την προηγούμενη απόφαση στην υπόθεση Google κατά Ισπανίας για τη μηχανή αναζήτησης μπορεί να βρουν ως ελεγκτές των δεδομένων. Και απάντησε το δικαστήριο ότι η επεξεργασία κάποιων κατηγοριών αφορούν όλους τους ε, ελεγκτές και τις μηχανές αναζήτησης και η ευαισθησία των δεδομένων είναι εκείνη που δικαιολογεί την καθολική και χωρίς εξαιρέσεις σε εφαρμογή αυτών. Ωστόσο αναγνώρισε το δικαστήριο ότι η ειδική επεξεργασία που έγινε από τη μηχανή αναζήτησης επηρεάζει την ευθύνη και τις υποχρεώσεις της μηχανής. Και κατέληξε ότι απαγορεύεται η επεξεργασία για λόγους διαγραφή συνδέσμου και μετά από επαλήθευση ε, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου προσώπου. Επίσης, κατέληξε το δικαστήριο ότι η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα διαγραφή συνδέσμων εκτός εάν διαπιστώνεται ότι εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 9 του GDPR και μπορεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να έχει δημοσιεύσει το ίδιο ε, τις πληροφορίες αυτές όταν ε, υπάρχει κρίσιμο δημόσιο συμφέρον στο να γίνουν γνωστά. Επίσης ε, ανέλησε το δικαστήριο το δικαίωμα στη λύθη και είπε ότι η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης αναφέρονται ρητά ως εξαιρέσεις στο δικαίωμα της λύθης. Επίσης η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο η συμπερίληψη του συνδέσμου είναι κρίσιμη για την προστασία της ελευθερίας πληροφόρησης, όπως ε, κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κανονικά, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων κυριαρχεί του δικαιώματος ε, της πληροφόρησης. Υπάρχουν εξαιρέσεις όμως ε, και σε ό,τι αφορά την προστασία της ζωής του προσώπου ε, ε, εξαρτάται όμως από το ρόλο του προσώπου αυτό, αν είναι δημόσιο πρόσωπο ή όχι. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά ε, τις ποινικέ διώξεις και καταδίκες και ορίζει το δικαστήριο ότι οι προφορίες που έχουν να κάνουν με κρεμίσεις υποθέσεις στη δικαιοσύνη και καταδίκες είναι δεδομένα που εμπίπτουν στο άρθρο 10 και τους αντίστοιχους ορισμούς του GDPR. Οπότε και η πληροφόρηση εμπίπτει σε αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση ζητήθηκε από τη μηχανή αναζήτησης να συμπεριλαμβάνει τους συνδέσμους αυτούς όταν ε, πρόκειται για λόγους ε, ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Και θύμισε εδώ την ομολογία του ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου και τόνισε τον ε, σημαντικό ρόλο που παίζει ο τύπος σε μια δημοκρατική κοινωνία και μεταξύ αυτών είναι αναφορές σε υποθέσεις της δικαιοσύνης. Ενδιαφέρεται το κοινό όχι μόνο, ε, ε, και έχει συμφέρον να ενημερώνεται για κάποιο επίκαιρο θέμα, αλλά το κοινό θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε αναζήτηση για παρελθούσες υποθέσεις. Ε, τέλος, θυμίζει το δικαστήριο ότι το δημόσιο συμφέρον σε ό,τι αφορά τις ποινικέ διαδικασίες διαφέρει σε βαθμό και μπορεί επίσης να αλλάζει ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Καταλήγει ότι η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να εκτιμά κάθε φορά την περίπτωση και αν ε, ε, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει να μην συνδέονται οι πληροφορίε αυτέ με το όνομά του. Εάν ε, ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να παραμείνει ο σύνδεσμος στο δικαστήριο, γιατί είναι ε, απαραίτητο απολύτως για να προστατεύονται χρήστε του διαδικτύου, τότε η μηχανή αναζήτηση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τα δικαιολογεί, α, μάλλον να, να προσαρμόζει τον κατάλογο των συνδέσμων όπως βγαίνει με το πιο πρόσφατο, πιο ψηλά στην ταξινόμηση της σελίδας. Και στην ίδια απόφαση το Συμβούλιο λέει ότι μια μηχανή αναζήτηση, όπως το Google είναι υποχρεωμένο να ε, συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις διατάξεις για κάποιες κατηγορίες δεδομένων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει πριν ζητηθεί ρητά από το ενδιαφερομένο πρόσωπο. Και καθώς οι μηχανές αναζήτησης ε, λαμβάνουν χώρα μόνο κατόπιν ε, τοποθέτησης των πληροφοριών από ένα τρίτο πρόσωπο, ε, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από αίτημα διαγραφής συνδέσμου. Θα πρέπει λοιπόν η μηχανή αναζήτηση να σταθμίζει πάντα το δικαίωμα στην προστασία τη ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Okay, thank you. Now we've got some room for discussion. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η παρουσίαση είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και βεβαίως και οι αποφάσεις οι ίδιες, οι υποθέσεις οι ίδιες είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ε, αποσαφηνίζουν κάποια στοιχεία τα οποία πολλοί έχουν συζητηθεί και έχουν συζητηθεί μάλιστα επί Μακρόν και στο ε, δικό μας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως στη δέσμη ε, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπου ε, προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε και να προωθήσουμε το δικαίωμα στη λύθη, το δικαίωμα στην διαγραφή στοιχείων τα οποία έχουν επιτευχθεί με παράνομο τρόπο ή στοιχεία τα οποία παραβιάζουν ε, καταφανώς ε, θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου ε, ή την ιδιωτικότητά του κλπ. Ε, κυρία Μπάρη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ίσως δεν το κατάλαβα καλά, αλλά είχα την αίσθηση ότι η πρώτη απόφαση ε, κερδίθηκε από την Google αλλά φαίνεται ότι ούτε αυτή δεν είναι ικανοποιημένη γιατί το δικαστήριο απεφάνθη ότι μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Αρχή να επέμβει και να τροποποιήσει τις αρχές χωρίς ε, το δικαίωμα να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Um, για διαγραφή δηλαδή από τους ε, καταλόγους ας πούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλες ερωτήσεις ρωτάει ο Πρόεδρος. I would, I would like the European Parliament Legal Service η νομική υπηρεσία του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα παρακαλώ ε, να αναφερθεί ε, στα θέματα αυτά, δηλαδή ότι για πρώτη φορά υπάρχει νομοθεσία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που όχι μόνο αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και καλύπτει και ένα νέο δικαίωμα το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα αυτό το δικαίωμα στην λύθη Δρουά Αλουμπλή Δερέτσο Αλολβίδο ο πρόεδρος αναφέρει την λέξη αυτή σε όλες τις γλώσσες. Για πρώτη φορά, για πρώτη πραγματικά φορά, Έχουμε αυτήν την δυνατότητα. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα διαγραφής κάποιων εικόνων, κάποιων στοιχείων ή οτιδήποτε άλλο. Με οποιαδήποτε μορφή στοιχείων τα οποία με κάποιο τρόπο ε, αποβαίνουν σε ζημία ενός συγκεκριμένου ατόμου και αυτό πραγματικά αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς, μακροτάτης μάχης που δώσαμε. Κυρία Ζήπελ, παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ. Αναρωτιόμουν αν πρέπει να υποβάλω το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι λαμβάνοντα υπόψη ε, αυτό το σχετικά νέο δικαίωμα, στην, στο δικαίωμα στη λύθη δηλαδή, αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτές οι αποφάσεις του δικαστηρίου έχουν ή δεν έχουν, ε, αποτε, δεν έχουν επίπτωση στο, στην ε, συνέχεια του GDPR. και βεβαίως ε, αυτή η δυνατότητα διαγραφής ε, θα πρέπει να γίνεται αναπερίπτωση μετά από εξέταση, θα εξαρτάται και από το άτομο μετά από εξέταση όλων των στοιχείων. Δεν αφορά μονάχα τα δικαίωμα του ατόμου και τα δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου, είναι και δικαίωμα των ατόμων απέναντι σε κάποια στοιχεία τα οποία άπτονται του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως το ερώτημα εδώ είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο ή ποιο άλλο όργανο θα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει ε, σταδιακά να δημιουργήσει έναν οδηγό σχετικά ε, με το ποια θα είναι τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην σχετική αυτή απόφαση. Δεν είμαι σίγουρη αν οι ίδιες οι αποφάσεις δίνουν ήδη κάποια στοιχεία, αλλά πάντως ε, οι υπηρεσίες προστασίας δεδομένων, οι υπηρεσίες της Κομισιόν, η νομική υπηρεσία έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται κάποια στοιχεία κοινού, ε, κοινής συνένεση ας πούμε, για το κατά πόσον το δικαίωμα στη λύθη ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να, ε, να ε, δοθεί σε περίπτωση που λόγοι δημοσίου συμφέροντος αντιτίθενται σε αυτή τη διαγραφή. Πρόεδρος, σχόλια. Legal service. Θέλετε να σχολιάσετε, παρακαλώ, να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Ναι. Ε, θα απαντήσω στα σχόλια. Όσον αφορά το πρώτο σχόλιο, κοιτάξτε, εξαρτάται από, ποια πλευρά βλέπει κανείς την απόφαση. Πάντως το δικαστήριο στην ουσία τεκμηριώνει ότι δεν υπάρχει κάτι στον κανονισμό που να δικαιολογεί την οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής του δικαιώματος στη λύθη εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το δικαίωμα αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο το δικαστήριο αναγνωρίζει ότι εάν έχει κανείς πρόσβαση στην, ε, στην πληροφορία από το εξωτερικό, αυτό πραγματικά μπορεί να έχει επίπτωση ε, στο ε, άτομο. Θα πρέπει να υπάρξει γενικότερα ένα υψηλό πλαίσιο προστασίας αλλά και σε αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να μελετήσουμε την έξω γεωγραφική ας πούμε διάσταση. Οι κανόνες ε, του GDPR είναι πολύ σαφείς. Μπορούμε να υποχρεώσουμε ε, στο, τον ε, πάροχο να διαγράψει όλα τα στοιχεία εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ε, εκτός αυτού υπάρχει και η εξισορρόπηση ανάμεσα ε, στα δικαιώματα του ατόμου και τα δικαιώματα του χρήστη του ίντερνετ και γι' αυτό ε, θα μπορούσε να υπάρξει μια υποχρέωση ε, για worldwide referencing, δηλαδή δικαίωμα στη λύθη παγκόσμιο. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από τις ε, ένομες τάξεις ε, των χωρών. Ε, επίσης, μην λησμονούμε ότι στην υπόθεση ε, Google κατά Ισπανίας δεν υπήρχε τότε ε, το δικαίωμα στην ελήθη. Αυτό το δικαίωμα θεσμοθετήθηκε μετά, στη διάρκεια της διαδικασίας. Και επίσης ε, ο νομοθέτης ε, προσπαθεί να παραμείνει ε, σε ισορροπία, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέχει το δικαίωμα του χρήστη του ίντερνετ και σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικότητας. Όσον αφορά τώρα την DPS, φαντάζομαι ότι μπορεί να δώσει κάποια ε, καθοδηγητικά στοιχεία όσον αφορά το άρθρο 17. Ε, πάντα όμως ε, στην προσπάθεια εξισορροπημένης λύσης και πάντα σε αναπερίπτωση αντιμετώπιση. Πρόεδρος, και εσείς θέλετε να υποβάλλετε κύριε Μπράιερ κάποια ερώτηση και μετά θα ακούσουμε ένα σχόλιο από την ε, Κομισιόν. Έχουμε εδώ εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου είναι ότι στο δικαίωμα στη το δικαστήριο αποφάσισε ότι η ισχύς ε, θα καλύπτει μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά την ίδια εβδομάδα το δικαστήριο πήρε μια απόφαση στην ε, περίπτωση ε, Κλάφιντ Μίτσιντα κατά του Facebook για τις αφαιρέσεις περιεχομένου και είπε ότι τα κράτη-μέλη, ε, μάλλον ε, όταν υπάρχει απόφαση, θα μπορούσε αυτή να έχει ισχύ παγκοσμίω ε, δυνάμει τη διεθνού νομοθεσία. Πώ μπορείτε να εξηγήσετε λοιπόν αυτή τη διαφορά, ή υπάρχει διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η σχετική διεθνή νομοθεσία θα λέει πάντοτε ότι τα, οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν μπορούν να έχουν παγκόσμια ισχύ. Ναι, πολύ χρήσιμη ερώτησή σας ε, και φυσικά όταν είχαμε την απόφαση για το Facebook ε, ξαφνικά είχαμε σχόλια ότι αποφάσισε διαφορετικά το δικαστήριο όμως πρέπει να πω εξ αρχής ότι από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της άποψη του δικαστηρίου δεν υπάρχει παρέκκληση. Τις ίδιες γραμμές ακολούθησε το δικαστήριο, την ίδια φιλοσοφία. Γιατί αν δείτε την απόφαση για το Facebook, το δικαστήριο έλαβε υπόψη την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αν δούμε τη διατύπωση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι ακριβώς ε, η ίδια, που είχε το δικαστήριο και στην υπόθεση Google και αν δούμε και τη διατύπωση του GDPR, το δικαστήριο λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα στην οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου ε, που θα εμπόδιζε αντίκτυπο παγκοσμίω. Έτσι λοιπόν παραπέμπει και πάλι στην εθνική νομοθεσία, δηλαδή και στην ε, υπόθεση Google το ίδιο έκανε το δικαστήριο, είπε. Δεν μπορούμε να το περιορίσουμε μόνο στα κράτη-μέλη, γιατί έχουμε ένα κανονισμό που θέτει τα κοινά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν βασικά εφαρμόζεται το δικαίωμα μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως το Facebook είπαν ότι δεν υπάρχουν κοινοί κανόνε ε, για τη δυσφήμιση. Διέπεται από τη διεθνή νομοθεσία, από διεθνεί κανόνες. Α το αφήσουμε αυτό λοιπόν στο διεθνές δίκαιο. Γιατί υπάρχει και το θέμα της σύγκρουσης δικαίων και εξαρτάται τι λένε αυτά τα δίκαια. Αν η Εθνική Αρχή μπορεί να ε, εκδώσει μια ε, εντολή που να ισχύει παγκόσμια ή όχι. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε τον ίδιο Γενικό Εισαγγελέα που πρότεινε την γνωμοδότηση και φυσικά απάντησε ε, σε αυτό το θέμα σε σχέση και με την υπόθεση της Google. Δηλαδή ουσιαστικά ακολουθεί την ίδια γραμμή το δικαστήριο. Δεν υπάρχει απόκληση μεταξύ των δύο αποφάσεων. Let's hear now. ακούσουμε τώρα τον ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, Φαρλίνα Μογιατόβιτς, ε, από την προστασία προσωπικών δεδομένων, το σχετικό τμήμα της Κομισιόν. Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμπληρώσω τις ε, δηλώσεις και την ερμηνεία της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Έχοντα κατά νου κάποιε από τι ερωτήσει που τέθηκαν εδώ, νομίζω ότι είναι και πάλι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν μιλάμε για διαγραφή των υποκείμενων πληροφοριών. Ήδη αυτό ίσχυε στην πρώτη υπόθεση Google, όπου η Λαβανγκουάρντια δημοσίευσε μία πληροφορία και η πληροφορία στη Λαβαγουάρδια παραμένει. Αυτό που αφαιρείται είναι μόνο ο σύνδεσμος προς αυτή την πληροφορία στο διαδίκτυο. Εδώ λοιπόν απαντώ και στην ερώτηση της κυρία Σίπελ σε σχέση με το θέμα της ισορροπίας ε, και του κοινωνικού συμφέροντος και τα νέα στοιχεία που έρχονται μετά το GDPR στις αποφάσεις Google 2, Google 3 είναι οι αναφορές που ε, χρησιμοποιούνται στο GDPR ε, στην καταχώρηση των πληροφοριών και αυτά που έχουμε τώρα στο άρθρο 17 του GDPR, το δικαίωμα στη διαγραφή, το δικαίωμα στη λύθη, ρητά. Κάτι που δεν ισχύει στην οδηγία. Λέει λοιπόν το δικαστήριο, είναι πολύ σημαντικό το διαδίκτυο για τη διάδοση των πληροφοριών. Δεν διαγράφω το παρελθόν γιατί όπου το είχαμε στη Λαβαργουάρδια, στην πηγή, ε, και όπου δημοσιεύτηκε αυτό παραμένει ως πληροφορία, αλλά αυτό που πρέπει να εξετάσω είναι σε ποιο βαθμό η διάδοση αυτής της πληροφορίας μπορεί να περιοριστεί σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν ένα άτομο λέει ότι αυτό πάει πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν υπάρχει ισορροπία. Τώρα, επιπρόσθετα σε αυτό που έγινε στην υπόθεση Google με ένα πιο ισχυρό στοιχείο της ελευθερίας του λόγου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση. Αν η Google κέρδισε τα πάντα, δεν είναι η θέση της Κομισιόν αυτή. Γιατί αν και η πρακτική της Google ήταν ε, ήδη να προβαίνει σε διαγραφή συνδέσμων ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Google ήθελε να το κάνει μόνο σε επίπεδο κράτους μέλους όπου είχαμε την προσφυγή του υποκειμένου. Και θα αναφέρθω εδώ στην τελευταίο ερώτηση που το πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε το Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων και πόσο μακριά μπορούμε να πάμε χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα αν έχουμε εξοδευτική εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, στον κανονισμό όπου έχουμε εναρμόνιση και έχουμε ευρωπαϊκό νόμο που εναρμονίζει το δικαίωμα το οποίο επικαλούνται τα άτομα ενώπιον του δικαστηρίου. Τα δικαστήρια λένε δεν έχουμε τίποτα και δεν μας το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε τέτοια περίπτωση να εφαρμόσουμε έξω εδαφικά τον GDPR. Και εδώ έγκυται η όλη συζήτηση για τους διάφορους βαθμούς προστασίας ε, του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης ε, παγκοσμίω. Η αυστριακή περίπτωση είχε να κάνει με την εθνική νομοθεσία και μας είπε το δικαστήριο εκεί ότι η εθνική νομοθεσία θα ελέγξει σε ποιο βαθμό δεν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς ε, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου σε ό,τι αφορά τι κατευθυντήριε γραμμέ. Οι κατευθυντήριε γραμμέ, σύμφωνα με το GDPR, ε, δεν παράγονται από ε, ή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασία των Δεδομένων ε, και υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την ε, εφαρμογή του δικαιώματος στη λύθη και υπάρχει πριν από το GDPR, δηλαδή είχε παραχθεί από την οδηγία μετά την πρώτη απόφαση για την Google και από ε, το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Έτσι λοιπόν όλες οι ευρωπαϊκές αρχές εργάζονται για την αναθεώρηση αυτών των κατηδίων γραμμών υπό το φως των δύο τελευταίων αποφάσεων του δικαστηρίου. Νομίζω ότι μέχρι τώρα κάλυψα όλα τα σημεία. για να συμπληρώσω τη δήλωσή σα, Παρακαλώ, αν μπορώ να βοηθήσω περαιτέρω, να μου το πείτε. Α, και μία προσθήκη. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ήθελα ότι η κυρία Μπάρλε ήθελε να αντιδράσει. Τελειώνεται. Ναι, ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι πρόσθετο. Για την δυνατότητα αρχέ προστασία των δεδομένων μπορούν ωστόσο σε εξαιρετικές καταστάσεις να σταθμίσουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ή της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, γιατί αυτό αναφέρεται στο σημείο 17.2 της απόφασης το δικαστήριο. Βασίζεται σε δύο άλλες αποφάσεις στο να περιορίσει λίγο ε, της, το αιτιολογικό της γλώσσας αυτών των αποφάσεων. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η στάθμιση από την Εθνική Αρχή. Ενώ λέει ότι σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες ε, υποχρεώνω μηχανή αναζήτησης παγκοσμίω να προβεί σε διαγραφή, αν ε, το κάνει η Εθνική Αρχή Προστασίας των Δεδομένων, τότε αυτή η αρχή δεν μπορεί να αφήσει εκτός του πεδίου εφαρμογής την μονάδα ε, την ενότητα συγγνώμη, της ιδιωτικότητας και την ε, ενότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όπως δηλώνεται στις δύο αποφάσεις στις οποίες παραπέμπει το δικαστήριο στην απόφαση της Google όταν λέει ότι υπάρχει ακόμα αυτή η δυνατότητα. Έτσι λοιπόν ακόμη και αν οι εθνικές αρχές τις δεδομένων κατά εξαίρεση αποφασίσουν για παγκόσμια εφαρμογή παρόλα αυτά η αποτελεσματικότητα και περιοχή του ενωσιακού δικαίου δεν μπορεί να υποσκαφτεί. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Μπάρλεϊ. Θα πω καλύτερα γερμανικά γιατί θα έχουμε καλύτερη ακρίβεια. Ε, Ακριβώ για να συμπληρώσω αυτό. Αν κατάλαβα καλά, είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες οι δικοί μας ισχύουν μόνο για την Ευρώπη και κατ' εξαίρεση μπορούν ε, οι εθνικές αρχές να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό τι σημαίνει. Εάν εμείς νομοθετήσουμε για περισσότερα παιδεία ε, σε σχέση με το δικαίωμα στη λύθη, περιορίζουμε τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Και σε σχέση με τα παγκόσμια ισχύοντα. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει περίπτωση με δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων να δημιουργηθούν προβλήματα στα κράτη-μέλη. Άλλα σχόλια υπάρχουν. Κομισιόν. Δεν ξέρω αν η νομική υπηρεσία θέλει να απαντήσει. Θέλετε εσεί τελευταία, όπω προτιμάτε. Νομική υπηρεσία. Θέλετε να παρεμβείτε στο σχόλιο της κυρίας Μπάρλεϊ. Ένα σχόλιο θα μπορούσε να είναι ότι οποιασδήποτε προϋποθέσεις ε, και αυτά όσο πιο πολλές είναι αυτές στον ε, ε, κανονισμό τόσο λιγότερη δυνατότητα απόκλησης μπορεί να υπάρχει. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν όμως θέλει να απαντήσει με πιο σαφή τρόπο. Κομισιόν. Κοιτάξτε, αυτός είναι κανονισμός. Ε, εμείς έχουμε πλήρως εναρμονίσει το δικαίωμα στη διαγραφή και το δικαίωμα στην λύθη, όπως ε, ε, αναφέρεται συχνά, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, το GDPR προσδίδει έναν συνολικό μηχανισμό συνοχής που με ομοιογενή και συνεκτικό τρόπο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ε, data authorities που είναι ε, οι επιβολείς και οι ελεγκτές ε, μπορούν να μειώσουν το περιθώριο ελιγμών που έχουν. Αν κατάλαβα καλά όμως, ο προβληματισμός σας είναι ο εξής. Αν προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα, τότε θα μειωθεί η δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας. Δεν νομίζω ή μάλλον δεν κατανοώ εάν ε, βάλετε περισσότερες ε, προϋποθέσεις πώς και με ποιο τρόπο το δικαίωμα ε, στην λύθη θα εφαρμοστεί βάσει του άρθρου 17 του GDPR. Ας πούμε, θα μπορούσατε να ε, ε, βάλετε περισσότερες εξαιρέσεις. Τότε θα σχηματοποιηθεί διαφορετικά ε, το, το δικαίωμα έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει προσφυγή ενώπιον των εθνικών αρχών, δικαστικών αρχών κλπ. Και επιπλέον εξαιρέσει θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Εάν όμως η ερώτησή σας αφορά περισσότερο την γεωγραφική ε, ε, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής ε, τότε από τη στιγμή που εφαρμόζεται ο ε, ενωσιακός νόμος δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν εφαρμόζεται μόνο στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικότητας αλλά και στις συγχωνεύσεις και τις αποσπάσεις κλπ. Α, και στην ευτυχία των ζώων. Στο σημείο 57 γίνεται αναφορά στην άμεση επίπτωση σε άτομο το οποίο βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα ισχύει το, ε, και εφαρμόζεται το δικαίωμα, αλλά θα πρέπει ε, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, να το διασυδέσουμε με ε, κάτι που αφορά το, την, εσωτερική, την ενωσιακή ένωμη τάξη. Είτε είναι δίκαιο ανταγωνισμού, είτε είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω εάν απήντησα στην ερώτησή σας, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να με βοηθήσετε λίγο για να καταλάβω ακριβώς τι ζητάτε. Δεν νομίζω, λέει ο Πρόεδρος, ε, ε, νομίζω ότι αρκετά μέχρι τώρα με αυτό το σημείο ε, και θα φτάσουμε στο θέμα το οποίο είναι το τελευταίο μας θέμα, 11.30 με 12.30, κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, συγγνώμη, με την ΕΚΟΝ. Ε, και ε, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, εξίσου σημαντικό με αυτά που είδαμε μέχρι τώρα. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσουμε την κοινή συνεδρίαση με την ΕΚΟΝ. if you will, we have one hour to go for an important point. Έχουμε ακόμα μία ώρα. Όχι βέβαια λιγότερο σημαντικά τα θέματά μας. Από το προηγούμενο έχουμε κοινή συζήτηση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Έχουμε πέντε σημεία στην ημερήσια διάταξη που τα έχουμε συμφωνεύσει σε ένα. Θα δούμε την ανακοίνωση Επιτροπή προ το Κοινοβούλιο και το Σύμβουλιο για την καλύτερη εφαρμογή του νοσικού πλαισίου για την κατηπολέμηση των εσόδων παράνομε δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Επίση, έχουμε την έκθεση τη Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Σύμβουλιο για την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά, η νομιμοποίηση εσόδων παράνομε δραστηριότητε και χρηματοδότηση τρομοκρατία που συνδέονται με διασυνορικέ δραστηριότητε. έκθεση Επιτροπή προ το Κοινοβούλιο για την εξολόγηση του πλατείου συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. FIU. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη διασύνδεση των εθνικών κεντρικών αυτοματοποιημένων μηχανισμών των κρατών μελών για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και έκθεση Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση των πρόσφατων υπόθεση ονικαζόμενη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε με την εμπλοκή δικαστικών ιδρυμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικεντρωθούμε τώρα στην ανακοίνωση της Κομισιόν της 24 Ιουλίου 2019 για το πακέτο για την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ε, για την καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου για την καταπολέμηση νομιμοποίηση εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Και όλα βασίζονται στην οδηγία για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η τέταρτη οδηγία που παρουσιάστηκε βάσει των συμπερισμάτων του Συμβουλίου για το Σχέδιο Δράσης ε, του Δεκεμβρίου 2018. Όπως ε, θα θυμάστε, αυτή η οδηγία αποτελεί κοινή αρμοδιότητα και της ΛΥΜΠΕ και της ΕΚΟΝ. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τα μέλη της ΕΚΟΝ που θέλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Πριν να ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι δυστυχώς αφού έληξε η η ε, ημερομηνία για τη μεταφορά στο ιστορικό δίκαιο τη τέταρτη οδηγία για το ξέπλυμα κρίματο. έχουν ξεκινήσει τη δικασία υπερβάση κατά διάφορων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ημερομηνία για τη μεταφορά τη πέμπτη οδηγία πλησιάζει. Είναι τον Ιανουάριο του 2020 και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εφαρμογής των οδηγιών από αρκετά κράτη-μέλη. Στην ανακοίνωση η Κομισιόν προτείνει ως ε, μία από τις ε, δυνατότητες για περαιτέρω εναρμόνιση του νομικού πλαισίου η οδηγία να γίνει κανονισμός και δεύτερον να, δοθεί, να δοθούν ε, ίσως κάποιες κάποια καθήκοντα εποπτείας συγκεκριμένα για την νομοποίηση παραμεσόδων, σε ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα για την κατάσταση της εφαρμογής ε, της νομοθεσίας για την σε παράνομων εσόδων φέτος στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο το Σεπτέμβριο του 2019. Είχαμε τη συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια και στο ψήφισμα το Κοινοβούλιο καλεί την Κομισιόν να αξιολογήσει στο πλαίσιο της ε, απαιτούμενης μελέτης αντεκτύπου οποιαδήποτε ε, μελλοντική αναθεώρηση της νομοθεσίας ε, για το αν θα χρειάζεται κάποιος κανονισμός, αν θα είναι κατάλληλος κάποιος κανονισμός και αν συγκεκριμένο, συγκεκριμένος φορέας που θα έχει καθήκοντα να εξετάζει το θέμα της νομικής παράνομων εσόδων ε, θα πρέπει να συσταθεί. Αυτό συνυπεγράφει από πολλούς συντονιστές της ΛΥΜΠΗ μαζί με τους συντονιστές της ΕΚΟΝ. Αυτό το ψηφίσαμε στις 19, συγγνώμη, το Σεπτέμβριο του 19. Και τώρα, θα ακούσουμε τους εκπροσώπους του Κομισιόν. Καταρχήν θα ακούσουμε την κυρία Βασιλιάδου, που είναι αναπληρωτής διευθύντρια ε, της Δέλτα, Δικαιοσύνης της Κομισιόν και κατόπιν θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε πολιτική ομάδα και όποιο άλλο βουλευτή θέλει να σχολιάσει για ένα λεπτό. Να είστε έτοιμοι για να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση. Παρακαλώ, η κυρία Βασιλιάδου, καταρχήν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τις Επιτροπές Λίμπε και Έγκον για την σημερινή πρόσκληση προκειμένου να παρουσιάσουμε το πακέτο μας για την ομιμπήση παράδομα εσόδων. Ε, καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του ξεπλήματος βρονικού χρήματο ήταν προτεραιότητα για την Κομισιόν και θα είναι και για την επόμενη θητεία. Ε, στο πλαίσιο αυτό του Ιουλίου του 2019 εκδώσαμε τέσσερις εκθέσεις ε, που παρουσίασε ο Πρόεδρος. Είχαμε νόμιμες υποχρεώσεις για τις τρεις εκθέσεις και άλλη μία εκδόθηκε κατόπιν συμπερασμάτων του Συμβουλίου και σχετικού αιτήματο. Έχω 15 λεπτά για να παρουσιάσω τι εκθέσει αυτέ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε, αλλά ευχαρίστω κατόπιν να ακούσω τι ερωτήσει σα. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να ξεκινήσω με την έκθεση, με αυτό που λέμε, ε, της κινδύνου σε, παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε την προσέγγιση που λέμε ότι βασίζεται στους κινδύνους. Δηλαδή όλα ξεκινούν από το να κατανοήσουμε τον κίνδυνο σε διάφορα προϊόντα και τομείς και μετά λαμβάνουμε βήματα για να μετριάσουμε τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αλλάζουν, δεν μένουν οι ίδιοι, επομένως ε, κάθε δύο χρόνια κάνουμε αυτό το εγχείρημα και προσπαθούμε να δούμε ποιος είναι ο κίνδυνος στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Το πρώτο εγχείρημα έγινε το 2017 όταν αξιολογήσαμε 40 προϊόντα. Το νέο ναι, εγχείρημα ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και αξιολογήσαμε 47 προϊόντα. Αξιολογήσαμε 7 προϊόντα παραπάνω δηλαδή επειδή κατανοήσαμε ότι υπάρχουν ε, νέοι κίνδυνοι για την εσωτερική αγορά. Και να σας δώσω κάποια παραδείγματα αυτό προέρχεται από τα εικονικά νομίσματα ή τα κρυπτονομίσματα, πώς αποκαλούνται, από ε, κάποια καθεστώτα επενδύσεων, από ελεύθερους λιμένες, από τον τομέα του ποδοσφαίρου κτλ. Έτσι λοιπόν θέλουμε να παρακολουθούμε τους κινδύνους αυτό που κάνουμε σε κάθε τομέα βλέπουμε τους κινδύνους και την ε, ευπάθεια που υπάρχει ξεχωριστά για τη χρηματοδότηση τρομοκρατία και ξεχωριστά για την ομοποίηση παράνομων εσόδων. Αυτό που είδαμε είναι ότι οι κίνδυνοι επεκτείνονται σε διάφορους τομείς. Δεν μιλάμε μόνο για τράπεζες όπως πιστεύουν πολλοί. Και ο κύριος κίνδυνος που εντοπίσαμε σχετίζεται με τα μετρητά ε, και με τις επιχειρήσεις όπου χρησιμοποιούνται μετρητά, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εναλλαγές. Επίσης έχουμε κίνδυνο από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως δικηγόρους, συμβολιογράφους, λογιστές λοιπά. Ο τομέα των στοιχημάτων επίσης φαίνεται να ενέχει ιδιαίτερου κινδύνους. Μπορείτε να διαβάσετε όλα όσα θέλετε για τους κινδύνους ε, στην δημοσίευσή μας. Προσπαθήσαμε να βρούμε επίσης ποιες είναι οι οριζόντιες ευαλωτότητες, ε, δηλαδή τι συναντάμε σε διάφορους τομείς και η μεγαλύτερη ευαλωτότητα που έχουμε είναι η ανωνυμία των συναλλαγών, ε, δεύτερον το να εντοπίζουμε τους πραγματικούς δικαιούχους και τα άλλα σχετίζονται στη λειτουργία των αρμοδίων αρχών που είναι υπεύθυνε για την νομιμοποίηση παρανομεσόδων και έχουμε αδυναμία στην εποπτεία και η λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Και τώρα θα σας παρουσιάσω δύο άλλες εκθέσεις ε, που παρουσιάσαμε γιατί μπαίνουν σε λεπτομέρεια στο να αξιολογήσουν το πώς λειτουργούν οι βασικές αρμόδιες αρχές και ποια ζητήματα αντιμετωπίζουν. Θα ξεκινήσω λέγοντα δύο λόγια για την έκθεση για τη μονάδα χρηματο... τι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών, που είναι κάποιε από τι κύριε αρμόδιε αρχέ. Δυνάμει το άρθρο 65.2 τη Οδηγία για την Ομιλία σε Μεσόδων μας δόθηκε εντολή να υλοποιήσουμε έκθεση για να δούμε ποια είναι τα εμπόδια στη συνεργασία των ε, στη συνεργασία των μονάδων με μονάδες τρίτων χωρών και για το αν ε, υπάρχει δυνατότητα παιδί εφαρμογή να έχουμε συνεργασία και ένα μηχανισμό υποστήριξη για τις FIUs σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βρήκαμε πολλές ελλείψεις δυστυχώς θα τις ομαδοτοποιήσω έλλειψη ορθής εφαρμογή στην εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης ανακαλύψαμε ότι πολύ συχνά οι μονάδες δεν ε, αντελάσσουν πληροφορίες με άλλες μονάδες. Υπάρχει έλλειψη feedback για τις οντότητες ε, και ε, ουσιαστικά είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος για απαντήσεις στα κράτη-μέλη κατόπιν έχουμε προβλήματα τεχνολογίας των πληροφοριών. Γιατί έχουμε το FIU Unit στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τη δίκηση της Europol που δυσλειτουργεί σε μεγάλο βαθμό, καταραίει το σύστημα και πρέπει να κάνουμε κάτι. Αλλά η κακή του λειτουργία πλήττει τη δυνατότητα των μονάδων να ανταλλάξουν διασυνοριακά πληροφορίες. Ένα άλλο πρόβλημα που βρήκαμε είναι η έλλειψη επαρκού συναρμόνηση για τι δραστηριότητε των FIUs οδηγεί σε ιδιαίτερα αποκλίνουσες ε, συγγνώμη, προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη. Έχετε σε κάποια κράτη-μέλη μονάδες που απαντούν ε, σε αιτήματα σε 24 ώρε, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη σε ένα μήνα. Έτσι λοιπόν, αυτά δεν θέλουμε να τα βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, βρήκαμε και κάποια διαφορετικά προβλήματα Έχουμε ομάδα εμπειρογνωμόνων που λέγεται πλατφόρμα για τις FIUs. Εκεί συναντώνται όλες οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, κάνουν καλή δουλειά στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, αλλά δεν ε, έχουν νομικές αρμοδιότητες προκειμένου ε, να υιοθετήσουν νομικά δεσμευτικούς κανόνες για τις FIUs. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα γιατί εκδίδει κατά τη διάρκεια η πλατφόρμα, κάποιες ε, μονάδες τις σέβονται, κάποιες τις αγνοούν. Ε, υπάρχει λοιπόν έλλειψη νομικών δεσμευτικών κανόνων από αυτό το φορέα. Δεν θα περάσω στα συμπεράσματα γιατί θα το κάνω στο τέλος για όλες τις εκθέσεις. Αυτό για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πολλά προβλήματα. Κατόπιν είχαμε μία έκθεση, μία post-mortem έκθεση, γιατί έτσι ε, αναφέρθηκε και στην πρέσβη του Συμβουλίου, αλλά είχαμε έτοιμο από το Συμβούλιο να εξετάσουμε πρόσφατες υποθέσεις ε, ξεπλήματο και να δούμε τι δεν πήγε καλά. Εξετάσαμε 10 ε, υποθέσεις, την Danske Bank, την Deutsche Bank, την Ebel Bank, ING, Nordia, Pilatus, Stata Bank, τη Societe Generale και Verso Bank. Ε, επιλέξαμε αυτές ε, γιατί πραγματικά παρουσιάστηκαν πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν σχετικά πρόσφατες και ήταν σημαντικές για να εντοπίσουμε τα προβλήματα. Και είδαμε τι συνέβαινε στις τράπεζες, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και σε επίπεδο διάφορων ε, αρμοδίων αρχών που έπρεπε να διερευνήσουν αυτά τα ζητήματα. Στις τράπεζες, λοιπόν, βρήκαμε και πάλι πάρα πολλά προβλήματα προβλήματα σε σχέση με την έλλειψη συμμόρφωσης, έλλειψη δέουσης επιμέλειας, δεν ανέφεραν τα γεγονότα στις εφεγιούς, προβλήματα διαχείρισης, περιορισμένες εσωτερικές ε, έρευνες, ε, ευθύνες ε, των διευθυντών, επίσης προβλήματα για το επιχειρηματικό μοντέλο ή προδιάθεση για κίνδυνο. Επίσης είδαμε σε κάποιες τράπεζες ότι είχαν καταθέσεις μη κατοίκων και είχαν επιθετική τακτική στην προσέγγιση των πελατών. Επίσης εξετάσαμε τις αρμόδιες αρχές για να δούμε τι κάνουν οι αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπίσουν ε, αυτά τα ελλείμματα στις τράπεζες. Καταρχήν ε, είδαμε τις εποπτικές αρχές, ε, πολλά προβλήματα και εδώ πολύ ανησυχητικό είναι το θέμα των περιορισμένων, πόρων, των περιορισμένων πόρων. Σε κάποιες χώρε, δύο άνθρωποι είναι αρμόδιοι της εποπτείας ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού τομέα σε μια χώρα. Εντελώς ανεπαρκές. Δεν αρκούσε η εποπτεία λοιπόν. Επίσης ε, κάποιες χώρε έκαναν μόνο τέσσερις φορές το χρόνο εποπτεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όχι μόνο για τις τράπεζες, για τις υπηρεσίες πληρωμής, το χάρη βρήκαμε ότι κάποιοι επόπτες δεν είχαν την απαραίτητη εμπειρία. Τα πρόστιμα τα οποία επέβαλαν δεν ήταν αποτρεπτικά, πολύ μικρά πρόστιμα δηλαδή. Και επίσης ε, κάποιοι δίσταζαν να επιβάλλουν και κυρώσει Σε μια χώρα βρήκαμε ότι δεν είχαν ποτέ επιβληθεί κυρώσεις. και πολύ η εικόνα λοιπόν. Κατόπιν πήγαμε στου ε, στους προληπτικούς επόπτες ε, γιατί αυτοί είναι φυσικά υπεύθυνοι για προληπτική εποπτεία αλλά πρέπει να δούνε τις επιτυχίες, ε, τη προληπτικής υποπτίας που σχετίζονται με την ομοποίηση παράνομων εσόδων. Και αυτό σχετίζεται σε ομαδική υποπτία συγγνώμη, η ομήλων, σε θέματα εταιρική διακυβέρνησης και επίσης βρήκαμε πολλά προβλήματα. Το πρώτο ήταν ότι μας είπαν οι υπόπτες, ε, είχαμε τέτοια καθήκοντα ε, για την ομοποίηση περνάμενων εσόδων, δεν το ξέραμε καν. Πολύ σοβαρό. Στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών βρήκαμε λιγότερα προβλήματα γιατί οι μονάδες δεν λάμβαναν απλώς πληροφορίες από τις τράπεζες ε, σχετικά με τις διάφορες ε, υποθέσεις. Ρωτήσαμε τις ε, μονάδες, λάβατε πληροφορίες για υπόπτες συναλλαγές. Όχι, μας είπαν. Έτσι λοιπόν εκεί είχαμε μικρότερο ρόλο των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτά ήταν τα γενικά πορίσματα των τριών εκθέσεων. Επειδή πρόκειται για μια μικρή έκθεση, αλλά είναι και πολύ σημαντική τελική έκθεση που αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο, ήταν μια έκθεση που σχετίζεται με την διασύνδεση των κεντρικών μητρών ή των τραπεζών. Η πέμπτη οδηγία υποχρεώ τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν κεντρικά μητρώα στις τράπεζες και η ίδια οδηγία ζητά από την Κομισιόν να δει ποια θα μπορούσε, ποιες θα μπορούσε να είναι οι τεχνικές δυνατότητε για να αλληλοσυνδεθούν αυτά τα μητρώα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εξετάσαμε και είδαμε ότι η Κομισιόν έχει όλη την απαραίτητη τεχνολογία γιατί συχνά προβαίνουμε σε διάφορους τομείς, σε τέτοιες διασυνδέσεις, ε, ε, εταιρικά, μητρώα, αφαιρεγγιότητα κτλ. Είναι λοιπόν εφικτό, έχουμε τη τεχνολογία, όμως τι μας λείπει, η νομική βάση για την διασύνδεση αυτή, γιατί δεν υπάρχει στην οδηγία αν ε, πρέπει να υπάρχει διασύνδεση, χρειαζόμαστε και τη νομική βάση. Τώρα θα πω κάτι γιατί είναι σημαντικό και δεν θέλω φυσικά να υποβαθμίσω τη σοβαρότητα των πορισμάτων, αλλά όλα αυτά τα πορίσματα ε, έλαβαν χώρα όταν ίσχυαν η τρίτη και τέταρτη οδηγία. Ε, και όπως ξέρουμε, ήδη έχουμε την πέμπτη οδηγία που θα τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να μεταφερθεί στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τον Ιανουάριο του 20. Και όχι μόνο αυτό, θα έχουμε την πέμπτη οδηγία, Έχουμε και την CRT5, τη CRT5 όπως την αποκαλούμε που άρει πολλά εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ των ε, εποπτικών αρχών. Έχουμε την αναθεώρηση που δίνει πολλές ε, εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τροπεζών ε, για το θέμα της νομοποίησης παρανομής Δεν Έχουμε την οδηγία για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα ενδυναμώσει τι συνεργασίε μεταξύ των δεκτικών αρχών και των FIUs. Έτσι λοιπόν πολλά μέσα θα τεθούν σε ισχύ πολύ σύντομα και θα ενισχύσουν σημαντικά το νομικό πλαίσιο. Το άλλο που θέλω να πω ότι ε, όλοι ανησυχούν και τα κράτη-μέλη αλλά και υποχρέες οντότητες αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι μια μεγάλη μετακίνηση προς βελτιώσεις το τελευταίο έτος. Βλέπουμε ότι πολύ περισσότεροι πορεί δίνονται στις αρμόδιες αρχές, ότι τροποποιούνται οι διαδικασίες, έχουν εργαλεία πληροφορικής για την επεξεργασία των πληροφοριών και όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε πολύ επιθετική ε, πολιτική διαδικασία σε παραβάση για την πρώτη οδηγία και καθώς ε, κρεμούν αυτές οι διαδικασίες επί είχαμε και επιτυχίες. Δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη έλαβαν βήματα για να θετήσουν νέα νομοθεσία για να κλείσουν τα κενά. Είμαστε εντελώς πεπισμένοι. Όχι. Αλλά παραμένουν μικρά ζητήματα σε σχέση με την εικόνα που είχαμε το 2017. Έτσι λοιπόν και αυτό λειτουργεί. Ναι, λοιπόν, ε, είναι κάπως ζωφερή εικόνα στις εκθέσεις, αλλά πολλά έχουν γίνει το τελευταίο έτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα κράτη-μέλη, από τα πιστοτικά ιδρύματα. Να πω όμως ότι στις εκθέσεις μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εντάξει, έχουμε αυτά τα κενά, έχουμε τις νέους νόμους, Έχουμε όλη αυτή την ευαισθητοποίηση των κρατών μελών που κάνουν βήματα. Είμαστε τώρα εντάξει, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στην νομοθεσία. Και η απάντηση είναι ναι. Η νομοθεσία πιθανότατα θα ε, χρήζε να καλυφθεί με λεπτομεριστήρους κανόνε και σε ό,τι αφορά τι αποπτικέ αρχέ και τι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών αλλά και τι υποχρεώσει για τι υποχρεώσει οντότητε. Να σα ε, δώσω δύο παραδείγματα. Η οδηγία λέει φαγιού εγκαίρω πρέπει να αντελάσει πληροφορίες. Αν δεν έχουμε συγκεκριμένε προθεσμίες, αυτό το θέμα πάντα θα είναι ανοιχτό. Κατόπιν, λέει η οδηγία. Σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επόπτες θα πρέπει να έχουν διευρυμένες αρμοδιότητες. Τι σημαίνει αυτό. Μπαίνουμε λοιπόν σε μία συζήτηση με τις αρχές. Αυτά που κάνετε αρκούν. Δεν ξέρω. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν βλέπουμε ότι η οδηγία θα πρέπει να καλυφθεί με περαιτέρω λεπτομέρειε. Όρο κανονισμό μερικέ φορέ χρησιμοποιείται γιατί να έχουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο εναρμόνιση. σω αυτό θα ήταν ένα κατάλληλο μέσο. Αλλά βέβαια δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι αποφάσει. Ένα άλλο γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι βλέπουμε κάποια ανάγκη για κάποια καθήκοντα να ανατεθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σχετίζεται και με τι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αλλά και με την εποπτεία. Ποια θα έπρεπε να είναι αυτά τα καθήκοντα, ή πόσο μακριά πρέπει να πάνε, πόσο λεπτό μέρη θα πρέπει να είναι. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να αξιολογήσουμε στο εγγύ μέλλον. Για να δώσουμε συγκεκριμένε απαντήσει και λύσει. Είδαμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, όπου δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο. Φαίνεται να υποστηρίζει την έκθεση και τις ιδέες μας για τη διόρθωση των προβλημάτων. Επίσης, ε, ίσως γνωρίζετε ότι υπάρχουν συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο ΚΟΦΗΝ ε, γενικά φαίνεται να υπάρχει γενική υποστήριξη και θα έχουμε συμπεράσματα το Δεκέμβριο. Έτσι λοιπόν χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι οι συνομοθέτες φαίνεται πρίμα φάση να υποστηρίζουν αυτές τις ε, περαιτέρω δεσμεύσεις. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Και εντός του χρόνου σας, ακούμε τώρα τα μέλη με τη σειρά των πολιτικών ομάδων. Από το ΕΛΚ, ο Αντιπρόεδρος Επιτροπής μας, ο κύριος Ράντεφ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Δεν ε, χωρά καμία βιβολία ότι συνέχεια έχουμε νέους κινδύνους και απειλές, εγκληματίες και τρομοκράτες που αναζητούν χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ξέπλυμα χρήματος. Η πέμπτη οδηγία ε, έρχεται να ενημερώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να την ευθυγραμμίσει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν, να ενσωματώσουν και να εφαρμόζουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οποιαδήποτε κενά ελλείμματα ή παραθυράκια σε πολλά κράτη-μέλη εκθέτουν σε απειλές και κινδύνους και τρομοκρατία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάλυση του κινδύνου επισημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι σε ανώνυμα προϊόντα όταν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος ή νέα προϊόντα όπως είναι τα κρυπτονομίσματα και τα εικονικά νομίσματα. Αυτοί οι κίνδυνοι ε, θα ξεπεραστούν εν μέρη όταν ενσωματωθεί η πέμπτη οδηγία για την νομιμοποίηση. Αλλά παραμένουν οι προκλήσεις και τα προβλήματα. Τα νέα προϊόντα κινδύνου, τα οποία έχουν εντοπιστεί, ε, συμπεριλαμβάνουν και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιοι ε, θα πρέπει να δηλώνουν ύποπτες συναλλαγές και ποιες θα είναι οι απαιτήσει ε, για την τήρηση της συμφωνίας σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Στα πλαίσια αυτά θα ήθελα να κάνω τις εξής ερωτήσεις δεν είναι σωστό να σκεφτούμε μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση που να καλύπτει και άλλα αθλήματα. Υπάρχουν επενδυτές από τρίτες χώρες ε, ε, που επενδύουν στον αθλητισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να ενημερώσει τη νομοθεσία για το ξέπλυμα και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επόμενη ερώτηση οι μονάδες ε, ε, οικονομικών πληροφοριών ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Υπάρχει μια έκθεση για το πλαίσιο συνεργασίας που τονίζει ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των FIU. Αλλά ως αποτέλεσμα του διαφορετικού νομικού καθεστώτος ε, οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και αρμοδιοτήτων τους, ε, ορισμένες από αυτές τις μονάδες δεν ε, μαθαίνουν καν τις προφορίες αυτές και πόσο μάλλον να τις ανταλλάξουν. Και επίσης είναι το θέμα της ανταλλαγής προφοριών με τρίτες χώρες. Τι προτίθεται λοιπόν να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχυθεί ο μηχανισμός συντονισμού και υποστήριξης. Υπάρχει η τράπεζα ε, Πιλάτου στην Μάλτα ε, που είναι πάρα πολύ ε, αμφισβητούμενη περίπτωση και αμφιλεγόμενη. Εσείς έχετε καμία επικοινωνία με τις μαλτεζικές αρχές για αυτό το θέμα. Η κυρία Σίπελα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ω συντονίστρια τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, θα ήθελα καταρχά να εκφράσω την ευγνωμοσύνη τη ομάδα μου για τη συνεχή εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το κρίσιμο θέμα του ξεπλήματο ε, χρήματο και τη καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Σα ευχαριστώ για τη σημερινή παρουσίαση. Όλα αυτά ε, τα έγγραφα και η δική σα παρουσίαση σήμερα δείχνουν ότι είναι πολλά τα κρίσιμα θέματα που απομένουν και θα πρέπει από κοινού να ε, ε, αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το θέμα του διεθνούς εγκλήματος που είναι και ε, ύπουλο. Από το Σεπτέμβριο είδαμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να σταθώ σε μερικά θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη δική μου πολιτική ομάδα. Στην ανακοίνωσή σας για την εφαρμογή του πλαισίου για το ξέπλυμα είναι πραγματικά ανησυχητική. Και στα 28 κράτη-μέλη, από ό,τι βλέπω, ε, έχετε ε, διαδικασίες επί σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, της οδηγίας, της τέταρτης, ε, που τον Ιούνιο του 2017 έλεγε η προθεσμία. Τώρα για την πέμπτη οδηγία λήγει η προθεσμία σε λιγότερο από δύο μήνες. Οπότε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι γίνεται, έχει αλλάξει η κατάσταση από τον Ιούνιο, έχει βελτιωθεί υπάρχουν περισσότερα κράτη-μέλη που μετέφεραν, ενσωμάτωσαν σωστά την οδηγία και έχετε καμία πληροφόρηση για το, τα πόσο θα τηρηθεί η προθεσμία το Ιανουάριο του 2020 για την πέμπτη οδηγία. Η έκθεση για την συνεργασία αναφερθήκατε στις μονάδες FIU. Υπάρχουν προβλήματα. Όπως ίσως γνωρίζετε, η ομάδα S&D εξακολουθεί να ζητεί ε, πανευρωπαϊκή FIU μια μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ξεπεραστούν πολλά προβλήματα που αναφέρει η εκθεσή σας. Ε, ε, μιλήσατε για το Συμβούλιο, αλλά θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες αν πραγματικά ε, είναι πιο θετική απόκριση τώρα του Συμβουλίου σε αυτή την ιδέα. Τι λένε τα κράτη-μέλη τώρα που έχουμε καταλάβει ότι η τρέχουσα συνεργασία χωλαίνει και δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της ανακοίνωσης ότι η μονάδα που ε, ασχολείται με το ξέπλυμα θα φύγει από την Γενική Διεύθυνση Just της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πάει στη Γενική Διεύθυνση FISMA. Αυτό τι σημαίνει θα ξεφύγουμε από τον ποινικό χαρακτήρα του ξεπλήματος και ε, ε, γιατί εμείς έχουμε και λόγο εκεί σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και την πληροφόρησή μας. Κύριε Νετσβέλτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν ε, για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα στο θέμα αυτό, στην προσπάθεια να καλύψει και κενά στην νομοθεσία, αλλά και κενά στην εφαρμογή και την επιβολή. Υπάρχει δεν υπάρχει δυνατότητα εξέβρεσης ε, της ε, διασύνδεσης, ε, δεν υπάρχει νομική βάση. Αναρωτιέμαι όμως γιατί η Κομισιόν δεν έκανε κάποια αντίστοιχη πρόταση, γιατί σε άλλες περιπτώσεις κινείται πολύ, κινείται πολύ γρήγορα έτσι ώστε να προτείνει κάποια τέτοια νομικό βάση. Γιατί διστάζει εδώ θα μπορούσε να υπάρχει διασύνδεση σε σχέση με το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με χρήματα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, ε, φορολόγηση κλπ. αποτελεί η δική τους αποκλειστική αρμοδιότητα. Α, όμως η Κομισιόν είναι ε, ανεξάρτητη και επομένως θα έπρεπε να προχωρήσει άσχετα από το τι πιστεύουν τα κράτη-μέλη. Θεωρεί η Κομισιόν ότι θα μπορούσε να προτείνει έναν ενιαίο ε, ελεγκτή γιατί η επιτήρηση με διάφορους φορείς ε, ε, είναι προβληματικός και ε, με αυτόν τον τρόπο εξασθενεί ιδιαίτερα η δυνατότητα επιβολής. όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, θεωρείτε ότι ασκεί πλήρως τον ρόλο της, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σκληρή. Τέλος, στην αρχή της παρέμβασής σας αναφερθήκατε στα χρυσά διαβατήρια, τις χρυσές θεωρήσεις σε βίζα από... Υπάρχει τέτοια νομοθεσία παντού, ε, αλλά παρόλα αυτά εμείς στρώνουμε τα κόκκινα χαλιά έτσι ώστε χρήματα τα οποία έχουν κερδιθεί μέσα από εγκληματικές πράξεις ε, να έρθουν εδώ ε, είναι λίγο σαν να έχουμε και το καρότο και το μαστίγιο μαζί και να μην χρησιμοποιούμε κανένα από τα δύο. και εν τέλει κάνουμε μια τρύπα στο νερό, όπως λέμε και στη γλώσσα μου. Ε, ε, πραγματικά έστω και αν η νομική βάση δεν είναι απόλυτα ισχυρή, δεν θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να προχωρήσει. Μήπως η Κομισιόν ε, ε θα έπρεπε απλώς να απαγορεύσει ε, τα χρυσά διαβατήρια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπρικμόντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε από την Επιτροπή. Ε, με χαρά βλέπει η ομάδα μου τα, ότι τα θέματα αυτά του ξεπλήματος και λοιπά παραμένουν σε ε, υψηλή προτεραιότητα ε, ε, και ελπίζουμε βεβαίως ότι και το ενδιαφέρον θα συνεχιστεί με την νέα σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα συμπεράσματα της ανακοίνωσης και τη θέση που έχει πάρει για τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερως χαιρετίζουμε τη βούλησή σας να κάνετε πλέον κανονισμό, να μετατρέψετε την οδηγία σε κανονισμό όσον αφορά το ξέπλυμα ε, χρήματος. Δεύτερο σημείο, το, οι εθνικές αξιολογήσεις κινδύνου ε, που ε, έχουν επιβεβαιώσει τους φόβους σχετικά με τις χρυσές βίζες και τα χρυσά διαβατήρια. Κατά την έννοια αυτή, θα μπορούσατε να σκεφτείτε την πλήρη κατάργηση αυτών των πρακτικών. Επίσης το θέμα της πλημελούς εφαρμογής παραμένει ένα ζήτημα. Ας πούμε, 80% των εταιριών ε, δεν έχουν ακόμα υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο, ε, ενώ έχει παρέλθει ε, προπολού η προθεσμία. Επίσης ξέρουμε ότι έχετε ξεκινήσει μία ε, διαδικασία ε, έρευνας, μελέτης ε, των θεμάτων αυτών. Έχουμε κάποια, κάποιο χρονοδιάγραμμα. Επίσης θα προωθήσετε τη σκέψη όσον αφορά ένα νομοθετικό εργαλείο το οποίο θα εφαρμόσετε σύντομα. Η κυρία Κάνκο. Κοιτάξτε, ε, είναι διαρκής αυτή η προσπάθεια καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος και επομένως θα πρέπει ε, διαρκώς να εξελίσσεται η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τα τελευταία πέντε χρόνια επανειλημμένα ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές και καταλήξαμε σε κάποια κοινή νομοθεσία. Ωστόσο, η πλημελής και διαφορετική εφαρμογή των κανόνων έχουν ε, ε, σαν αποτέλεσμα να ε, υπάρχουν εξα... κοινά κενά ακόμη και βεβαίως να δυναμητίζεται η νόμιμη οικονομική δραστηριότητα στις χώρες μας. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε νέον κανονισμό. Έχουμε δύο χρόνια τώρα που έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και εντωμεταξύ το πρόβλημα μεγαλώνει θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να καταρτιστούν. Ε, ε, ας πούμε έχουμε το EDPS και το GDPR. Ε, χρειαζόμαστε μία αντίστοιχη νομοθεσία ή πρακτική η οποία θα οδηγεί στην αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα θέματα της ε, του ξεπλήματος ε, χρήματος ε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ έχει αποδειχθεί ότι καλύπτεται από τέτοιου είδους οικονομία. Πραγματική ασφάλεια χρειάζεται η οποία όμως δεν διασφαλίζεται μονάχα από την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Τρεις ερωτήσεις. Ε, η καλή υλοποίηση είναι σημαντικό θέμα, έστω και αν δεν είναι το πιο σημαντικό και καμιά φορά το ξεχνάμε. Η νέα Κομισιόν έχει διαρθρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ε, ε παρεμφερεί θέματα ε, μοιράζονται σε διαφορετικά χαρτοφυλάκια διαφορετικών επιτρόπων. Πώς μπορεί με αυτό το πλαίσιο να γίνει καλή συνεργασία. Ποια είναι τα, τα, τα πρακτικά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την καλή συνεργασία των ε, αρχών επιτήρησης ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Πώς πιστεύετε ότι ε, μπορεί η καλή συνεργασία να βελτιωθεί τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ η κυρία Κιούρη. For anyone? No. Όχι ΚΟΕ. Έλκ είμαι. Α, έλκυσαστε. Καλά. We'll take the Από την ΚΟΕ κανείς. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα μέλη. Και εσείς, κυρία Γκιόρη, από το ΕΛΚ. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν προτίθεμαι να αλλάξω πολιτική ομάδα. Ε, νομίζω ότι δεν είναι κανείς εδώ παρόν που θα ήταν κατά της επιτάχυνσης, κατά πολέμησης, χρηματοδότησης τρομοκρατίας και του ξεπλήματος. Θα πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε. Παρόλα αυτά, θα ήθελα κάτι να θυμίσω που είπαν και πολλοί συνάδελφοι. Ε, ε, βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαδικασία νομοθέτησης τα τελευταία χρόνια με την τέταρτη και πέμπτη οδηγία. Ακούσαμε ότι... Προθεσμία ε, για τη μεταφορά της πέμπτης οδηγίας εκπνέει σε δύο μήνες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία σχεδόν καθόλου για το πώς ε, δουλεύουν στην πράξη αυτές οι νέες νομοθεσίες και τι αντίκτυπο θα έχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό τον τόμο που εξέδωσε και δείχνει ότι ε, πραγματικά έχουμε ιστορία σε αυτό αυτή την υπόθεση και δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε γιατί δεν έχει τελειώσει καθόλου αυτή η υπόθεση. Απλώς θα πρότεινα να κατεβάσουμε λίγο τις προσδοκίες μας, να μην ζητάμε, μέχρι και οργανισμό ακούσαμε, ε, να ζητείτε στην ΕΚΟΝ στις αρχές Σεπτεμβρίου. Δεν χρειαζόμαστε τώρα νέα θεσμικά όργανα ή νέα μέτρα και νέα μέσα ε, για να καταποτελεμήσουμε κάτι ε, με το οποίο όλοι διαφωνούμε. Και να προσθέσω κάτι ακόμα. Ε, πιστεύω ότι εδώ είναι ένα κλασικό πεδίο όπου θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και να ε, έχουμε εμπιστοσύνη στους εθνικούς θεσμούς. Βεβαίως πάντα χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό είναι το τελευταίο Υπάρχουν πολλές πληροφορίες πάρα πολύ εμπιστευτικές που κυκλοφορούν όταν πρόκειται για χρηματοδότηση και προσπαθούμε να ελέγξουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν αυτό γίνεται μέσω ε, των κρατικών αρχών, είναι καλό και των αρμοδίων οικονομικών αρχών. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να δημιουργούμε νέους θεσμούς και νέους οργανισμούς, διαχέεται η πληροφορία και μπορεί να έρθουν σε πολύ δυσμενή θέση οι ίδιες μας οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά Ινστιτούτα. Existing actors. Thank you so much. Λοιπόν, μας φτάνουν οι οργανισμοί που έχουμε και καλύτερα να συνεργάζονται αυτοί μεταξύ τους, να μην δημιουργούμε νωρίς. Νομίζω ότι η κυρία Μετσόλα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, Let me also... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ε, καλωσορίσω τη σκληρή δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και οι συνάδελφοι. Περιμένουμε με χαρά να ακούσουμε όλες τις απαντήσεις. Έχω μια ερώτηση που βασίζεται σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για την Τράπεζα Πιλάτους στη Μάλτα και ε, τα χρυσά διαβατήρια και τις χρυσές θεωρήσεις. Τι είδαμε στη Μάλτα με την υπόθεση Πιλάτους. στα χαρτιά ήταν όλα καλά, αλλά όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες είχαν παρακαμφθεί. Και ήρθε και μεγάλη πολιτική στήριξη η τράπεζα. Αλλά αυτή η τράπεζα ήταν σκιώδης ε, ε, για να ε, προστατεύει επιλεγμένα πρόσωπα από τον έλεγχο. Και υπήρχαν άνθρωποι που αγόραζαν ευρωπαϊκά διαβατήρια, διαπλεκόμενοι με πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, και σταμάτησαν ε, όταν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε συνέλαβαν τον πρόεδρο της τράπεζας. Τι γίνεται λοιπόν όταν ε, είναι όλα εντάξει, ωραία και καλά στα χαρτιά, ενημερώνονται οι πάντες ότι κάτι τρέχει, αλλά δεν αναλαμβάνεται καμία δράση. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις εικονικές τράπεζες. για τα διαβατήρια. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κράτη-μέλη, όταν κάποιο αγοράζει ένα τέτοιο χρυσό διαβατήριο, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Χένια Λιώμα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο της και ταυτόχρονα μας ανησυχεί και μας θορυβεί να ακούμε ότι ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν πηγαίνουν καλά σε ό,τι αφορά τις χρηματικές ροές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση ε, με την αξιότιμη συνάδελφο του ΕΛΚ, προβληματίζομαι ως νέο μέλος εάν είναι σωστός τρόπος αυτό, αυτές οι οδηγίες. Γιατί και ο επιχειρηματικός ε, κόσμος ζητάει να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη για να μην χάνουν χρήμα και χρόνο μέχρι να μάθουν τις διάφορες κουλτούρες και τα ήθη και τα έθιμα στα διάφορα κράτη-μέλη. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να έχουμε ενδεχομένω πιο δεσμευτική ε, νομοθεσία και τους ίδιους κανόνες παντού. Και δεύτερη ερώτηση, όποτε μπορούμε ή μάλλον πώς μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρχή που να εγγυάται ότι κάθε κράτος μέλος κάνει τη δουλειά του. Γιατί αν υπάρχουν παραθυράκια στην νομοθεσία των κρατών μελών, τι να το κάνουμε αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριο Σκούκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσίαση και αυτό το πολύ βοηθητικό έγγραφο το και πραγματικά μου άρεσε περισσότερο το δεύτερο μισό, γιατί ως ε, πρώην εισαγγελέας νομίζω ότι ήξερα διάφορους τρόπους που γίνεται το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι εντοπίζεται διάφορα ε, διάφοροι κρυπτονομίσματα, ATM, δηλαδή παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους γίνεται η νομιμοποίηση και ποτέ τους έχω ξανακούσει. Και άλλο είναι που βλέπουμε λοιπόν ε, όλα αυτά να προσδιορίζονται. Αναρωτιέμαι πω ε, κάτι έχετε παραβλέψει πολιτικέ οργανώσει ε, που οδηγούν σε, στη δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα των εξωτερικών υποθέσεων και τη Δημοκρατία. Γιατί στη δική μου χώρα δεν εφαρμόζονται οι κανόνες για τις πολιτικές οργανώσεις. Δηλαδή και ενώ μια μικρή επιχείρηση πρέπει να ελέγξει από πού έρχονται τα ε, χρήματα. Πολιτικά κόμματα δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε και αυτό για να σταματήσουμε την τρομοκρατία και το έγκλημα, αλλά και να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα τη δημοκρατία μα. Και συμφωνώ με του συναδέλφου που λένε ότι πρέπει να έχουμε του ίδιου κανόνε σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν είναι μόνο σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα, αλλά ε, να είμαστε και δίκαιοι απέναντι στου ανθρώπου που έχουν μικρέ επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος βουλευτής να θέσει ερωτήματα ή ανησυχίες, τότε ας ξανακούσουμε την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Βασιλιάδου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Θα βάλω τα δυνατά μου να τις ομοδοποιήσω και να απαντήσω αλλά χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι ενδιαφέρεστε και έχετε και γνώση διάφορων πτυχών της δουλειά που κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχήν από το θέμα της εφαρμογής, γιατί πολύ θα ερωτήσει για αυτό το θέμα. Μία από τις ερωτήσεις είναι αν έχει υπάρξει πρόοδος από τον Ιούνιο. Έχει υπάρξει. Εμείς κλείσαμε τη δικασία υπέρβαση για τέσσερις χώρες τον προηγούμενο μήνα και σκοπεύουμε να το κάνουμε για άλλες τέσσερις χώρες αυτό το μήνα. Επίσης λάβαμε κοινοποίησεις από πολλά κράτη-μέλη για νέες νομοθεσίες που έχουν υιοθετήσει. Και ξέρετε, υπάρχει γραφή ερωτία στην Κομισιόν, πρέπει να τις μεταφράσουμε και να τις αξιολογήσουμε. Χρειάζεται χρόνος, όμως βλέπουμε να υπάρχει σημαντική πρόοδος. Επίσης, έλαβα μια ερώτηση για το αν περιμένουμε μια πέμπτη οδηγία να, η πέμπτη οδηγία να μεταφερθεί στο ιστορικό εγκαίος. Έξι ε, κράτη-μέλη μας έχουν κοινοποιήσει ότι έχουν μεταφέρει την οδηγία ήδη. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες κοινοποίησεις τους επόμενους δύο μήνες. Αλλά, όπως πάντα, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Ελπίζουμε όμως ότι μέχρι την Άνοιξη θα λάβουμε τις περισσότερες κοινοποίησεις που χρειαζόμαστε. Ακούσε επίσης κάποιες ερωτήσεις ε, για τη μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης και το χρονοδιάγραμμα. Πολύ από τη δουλειά που προέκυψε από τα Panama Papers ήταν πολύ χρήσιμη για μας. Και μάθαμε ότι δεν αρκεί να βλέπουμε την νομοθεσία των κρατών μελών, αλλά και πώς εφαρμόζουν το νόμο στην πράξη. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να προβεί σε αυτή τη μελέτη με επιτόπου ε, επισκέψεις και με ερωτηματολόγιο. Έχουμε 300 ερωτήσεις ε, για να σχηματίσουμε μια καλή εικόνα για το τι συμβαίνει επιτόπου. Μόλις ξεκίνησε η μελέτη αυτή, και θα εργαστούν μέχρι το 2021. Χρειάζεται χρόνο, γιατί θα πρέπει να επισκεφτούν όλα τα κράτη-μέλη. Και σκοπεύουμε να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα στην έκθεση που θα δημοσιεύσουμε βάσει του άρθρου 65 τη οδηγία το 2022. Χρονοτριβή κάπω, αλλά είναι κάτι πλήρες και θα γίνει ορθά. Ακούσαμε κάποια σχόλια που τόνισαν την ανάγκη καλή συμμετοχής και της παροχής βοήθειας στα κράτη-μέλη και να τα υποχρεώσουμε να υλοποιήσουν τα καθήκοντά τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μέσω τη αξιολόγηση κινδύνου είδαμε ότι είχαμε ένα μεγάλο κίνδυνο από του δικηγόρου και του συμβολογράφου. Κάναμε λοιπόν πέρσι κάποια κατάρτιση για τους συμβολογράφους σε όλη την Ευρώπη. Φέτος ε, θα την υλοποιήσουμε για τους νομικούς, ε, για να κατανοήσουν όλα τα καθήκοντα που πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Έτσι λοιπόν ε, εξετάζουμε το θέμα της κατάρτισης και να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της οδηγίας. Υπάρχει ένας φορέας στην Κομισιόν, RSS νομίζω λέγεται, δεν θυμάμαι ποτέ να σας εξηγήσω τα αρχικά, αλλά δίνει διαφορετική υποστήριξη στα κρατη για να εφαρμόσουν τους διάφορους κανόνες. Και όντως Παρέχουμε υποστηρίξη σε, πέντε συγγνώμη, σε 7 κρατημέλη πέρσι για θέματα νομοποίησης παρανομών εισόδων και φέτος λάβαμε αιτήσει από άλλα πέντε κράτη. Έτσι λοιπόν εργαζόμαστε και από αυτού. Για την Κομισιόν συμφωνεί μαζί σας ότι το πρώτο βήμα είναι η ορθή εφαρμογή των σημερινών κανόνων. Λάβαμε κάποιες ερωτήσεις για τα εμπόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διάφορων αρμοδιών αρχών. Άλλο είναι να μιλάμε για εμπόδια και η δική μου πρώτη αξιολόγηση είναι ότι κατόπιν της εφαρμογής της πέμπτης οδηγίας και όλων των άλλων που σας ανέφερα, των καινούριων, δεν θα υπάρχουν τόσο πολλά εμπόδια για τη συνεργασία. Όμως αυτό που λείπει είναι μια υποχρέωση συνεργασίας. Δηλαδή, ναι, άλλο είναι να πεις ε, σε μια αρχή μπορείς να ανταλλάξεις πληροφορίες και άλλο να τις πεις πρέπει να ανταλλάξεις πληροφορίες. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε λοιπόν στα επόμενα βήματα για να δούμε αν θα πρέπει να ενισχυθούν οι κανόνες. Λοιπόν, έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα για ένα EU-FIU ή όπως τον λέμε καλύτερα ένα μηχανισμό συντονισμού για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πήγα στην πλατφόρμα FAU για να παρουσιάσω τη σχετική έκθεση και πραγματικά τρομοκρατήθηκα. Αλλά μετά ήταν πολύ θετικά τα σχόλια που έλαβα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα από τις εφαγίους και τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Συμφωνούσαν με τα πορίσματά μας σε μεγάλο βαθμό και ένα τέτοιο μηχανισμός συντονισμού και στήριξης θα ήταν κάτι χρήσιμο. Έτσι λοιπόν μα καθησύχασα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτού. Ερωτήσεις ε, για μία εποπτική αρχή είναι κάτι που θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε. Το γράψαμε σε αυτή την έκθεση post-mortem. Βλέπουμε προσθεμένη αξία στο να αναθέσουμε κάποια θήκοντα σε ένα κεντρικό όργανο. Νομίζω ότι και ο κ. Ντομπρόφσκι τον έφερε στην ακρόασή του. Επομένω, ο νέο αρμόδιο αντιπρόεδρο φαίνεται ότι σκοπεύει να λάβει κάποια τέτοια μέτρα, τουλάχιστον να κάνει μια σοβαρή αξιολόγηση για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Τώρα για την τράπεζα πιλάτους ένα εκατομμύριο πράγματα πήγαν λάθος. Υπήρχαν όλοι οι κανόνες και οι κατάλληλοι φορείς, αλλά δεν ελήφθη ιδιαίτερη δράση. Για να συνδέσω την, τα όσα είπατε, μετά όσα είπε η κυρία Ίντβελ με το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών βρήκε ότι η Μαλτεζική μονάδα είχε παραβιάσει το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν ανέλαβε δράση, επειδή δεν παρακολούθησε την κατάσταση, δεν επόπτευσε τις δράσεις των ανθρώπων κτλ. Είδαμε ότι είχαμε στη συνέχεια γνωμοδότηση της Κομισιόν ε, που καλούσαν τις Μαλτεζικέ, τη Μαλτεζική Φεγιού να αλλάξουν ε, τη δράση τους ε, και Πρέπει να είμαι δίκαιη σε αυτήν την κατάσταση και να πω ότι η Μαλτεζική μονάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, μεγάλη βελτίωση για να εθετήσει τι διάφορε νομοθεσίε, ε, τα διάφορα εργαλεία, τεχνολογίε των πληροφοριών. Απλώ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πράξη, στην πρακτική εφαρμογή. Πρέπει να δούμε λοιπόν και την εφαρμογή των νόμων. Είμαστε σε στενή επαφή με του Μαλτέζου. Για τι χρυσέ θεωρήσει, δύσκολο αυτό το θέμα και δεν είναι ένα από αυτά τα θέματα που γνωρίζω καλύτερα. Εδώ εκπροσωπώ την Κομισιόν, δεν εργάζομαι επί του θέματος αυτού. Από όσο καταλαβαίνω, θα μπορούσαν να υπάρχουν νομικά εμπόδια, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, να ρυθμίσει η Κομισιόν ή να απαγορεύσει αυτές τις θεωρήσεις, αλλά σίγουρα ενδιαφέρει την Κομισιόν, γι' αυτό είχαμε νωρίτερα φέτος την έκθεση τουλάχιστον τι έχουμε ως προς ε, την νομοθεσία. Μία απέτηση στην οδηγία για την νομοποίηση παράνομων εισόδων ε, εκεί όπου έχουμε ε, κάποιες συναλλαγές που συνδέονται με ετούντες ε, τέτοιων χρυσών θεωρήσεων θα πρέπει να έχουμε κάποιους συνεχισμένους ελέγχους γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις αυτές ως ενδυνάμει επικίνδυνες. Τώρα, για τη διασύνδεση των κεντρικών μητρών των τραπεζών. Πρόκειψε από τις διαπραγματεύσεις της πέμπτης οδηγίας. Δεν ξέρω πώς κατέληξα εκεί. Δεν υπάρχει νομική βάση τώρα. Αλλά δεν ε, διστάζουμε, ούτε τεμπελιάζουμε. Σας διαβεβαιώ, το θέλουν τα κρατημέλη γιατί θα γλιτώσουν πάρα πολλά χρήματα με ένα κλικ να μπορεί να δει κανεί όλα τα μητρώα. Αλλά το στο μέλλον θα γίνει ε, ένα εγχείρημα για να αναφερθούν όλοι οι κανόνες, για να γίνει αυτό άπαξ με ένα και μόνο μέσο και όχι με πολλά ξεχωριστά νομοθετικά μέσα, αλλά αυτό θα γίνει όταν θα αναλάβει και η νέα Κομισιόν. Υπήρχε μια ερώτηση για το ποια μέρη της οδηγίας ε, μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο να μετατραπούν σε κανονισμό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο άχθος στον ιδιωτικό τομέα γιατί θα πρέπει να σεβαστεί πάρα πολλού διαφορετικού κανόνε. Γιατί όταν βλέπουμε τι απαιτήσει για τι υπόχρεε οντότητε, βλέπουμε πολλέ αποκλήσει στα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι που θέλουμε να εξετάσουμε. Πώ μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να άρουμε κάποιο από το άχθο τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βέβαια όλα όσα λέω, αυτά είναι πράγματα που θα εξετάσουμε. Δεν δεσμεύομαι σε τίποτα γιατί θα πρέπει να κάνουμε Καταλληλικές αξιολογήσεις, αλλά ήθελα να σας πω ποιο είναι το αρχικό μα σκεπτικό. Νομίζω ότι απάντησα στις γενικές ερωτήσεις, ίσως να μην τις απαντήσα όλες, αλλά μπορώ να παραμείνω και μετά τη συνεδρίες, αν θέλετε, ή αν θέλετε να στείλετε γραπτός ερωτήσεις και να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Αν δεν έχετε άλλα σχόλια, φτάνει για σήμερα. Έχουμε συνεδρίαση και το απόγευμα νωρίς ξεκινάμε, στις 2 η ώρα. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη. Ραντεβού στις 2 και σας ευχαριστώ.